καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και ένα μεγάλο τμήμα των νομοθετικών εργασιών του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή Περιβάλλοντο θέλει πολύ να προστατεύσει τι συνθήκε για την υγεία, την ισότητα τη πρόσβαση στην περίθαλψη για όλου του ασθενεί στην Ευρώπη και για τα μέγιστα επίπεδα ασφαλεία σε όλη την επισητιστική, στην, στην ε, αλυσίδα των τροφίμων. Είναι καρδιοχειρούργο αντρικάτη, έχει 20 χρόνια εμπειρία στον ιατρικό του τομέα στη Λιθουανία ήταν Υπουργό ε, Υγεία από το 2012 μέχρι το 2014, περίοδο κατά την οποία η Λιθουανία είχε και την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από, μετά τα 20 χρόνια κοινοβουλευτικής ε, εμπειρίας, διότι ήταν βουλευτής για 6 θητείες στο Λιθουανικό Κοινοβούλιο, πρόσθεσε και αυτή την εμπειρία, ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής για Ευρωπαϊκά Θέματα και ηγήθηκε τη λιθουανική αντιπροσωπεία για τη Σύμβαση για το Μέλλον της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε αυτή η ακρόαση διοργανώνεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος σαν καθήλυνα αρμόδια επιτροπή και την Επιτροπή Γεωργίας ε, που είναι συνδεμένη επιτροπή. Έχουμε 45 ομιλητές και 6 από την Επιτροπή Γεωργίας. Να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τις κατακτήριες γραμμές για την έγκριση των υποψηφίων Επιτρόπων αξιολογεί τους υποψήφιους επιτρόπους στο Κοινοβούλιο βάσει των γενικών τους ικανοτήτων, την αφοσίωσή του για τα ευρωπαϊκά θέματα και την ε, προσωπική τους εξαρτησία επαληθεύει κατά πόσο γνωρίζουν τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και τη δυνατότητα που έχουν όσον αφορά την επικοινωνία. Πριν από την ακρόαση, ο Επίτροπος απάντησε γραπτός στις ε, γραπτές ερωτήσεις που του θέσαμε οι απαντήσει στα αγγλικά διανεμήθησαν στου βουλευτέ στι 26 Σεπτεμβρίου και όλε οι άλλε γλωσσικέ εκδοχέ έχουν διανεμηθεί χτε το απόγευμα. Όσον αφορά τη δομή τη συζητήσεω, ο υποψήφιο επίτροπος θα κληθεί να προβεί σε μια εισαγωγική δήλωση που δεν θα κρατήσει πάνω από 10 λεπτά και μετά στο τέλος της συνεδριάσεως θα έχει ένα πεντάλεπτο στη θέση του τόσο ώστε να προβεί σε μια σύνοψη, σε καταληκτική δήλωση. Θα υπάρξει χρόνο για 45 ερωτήσει βουλευτών κατά τη διάρκεια τη ακρόαση. Σε τέσσερι ομάδε θα μοιραστούν ερωτήσει. Η πρώτη ομάδα θα αποτελείται από 7 μεγαλύτερε ερωτήσει, 5 λεπτού, με το σύστημα ping-pong που θα ακολουθήσουμε. Θα τεθούν ερωτήσει εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα έχουμε ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση, ένα λεπτό για συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό για συμπληρωματική απάντηση. Μετά θα υπάρξει δεύτερος γύρος, 26 συντόμων ερωτήσεων, τριών λεπτών συνολικά, που θα τεθούν από τα μέλη της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ένα λεπτό για την αρχική ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Και στον τρίτο γύρο όμως έχουμε συμπεριλάβει τις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Γεωργίας Ερωτήσεις σύντομες θα είναι αυτές και θα καταλήξουμε με 7 σύντομες ε, ερωτήσεις από την πλευρά των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Το τέλος λοιπόν, για, μάλλον για να ολοκληρώσουμε τη συνεδρία εγκαίρως, διότι προβλέπει να, θα πρέπει να διαρκέσει ακρόαση τρεις ώρες, για να είμαστε εγκαιροί καλούμε και τους συναδέλφους στον υποψήφιο επίτροπο να σεβαστούν τον χρόνο ομιλίας. Θα υπάρξουν 5 δευτερόλεπτα ανοχής για τους βουλευτές και 10 δευτερόλεπτα ανοχής για τον επίτροπο. Αν περάσουν αυτά, το μικρόφωνο θα κλείνει. Ένας αστερίσκος θα εμφανίζεται επί τη οθόνης 10 λεπτά, 10 συγγνώμη δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου ομιλίας και το σφυράκι του Προέδρου πάση περιπτώσει θα υπενθυμίζει ότι λύγει ο χρόνος. Υπενθυμίζω ότι η διαρμηνία προβλέπεται σε 23 γλώσσες. Συνεπώς όλοι οι ομιλητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα τους. Η συζήτηση επίσης μεταδίδεται και στο διαδίκτυο μέσω streaming στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και από εκεί θα μπορείτε να κατεβάσετε την ηχογράφηση της ακρόασης. Δίνω αμέσω το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο, τον κύριο Ανδρουκάητη, ούτω ώστε να προβεί στην αρχική του δήλωση. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νιώθω μεγάλη τιμή που ήσταμε σήμερα ενώπιόν σας ως τμήμα της ομάδος του Jean-Claude Juncker για την Επιτροπή ενώπιον των δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των λαών της Ευρώπης, ώστε να ανταλλάξω απόψη μαζί σας, να επιζητήσω την έγκρισή σας για τον διορισμό μου ως Ευρωπαϊκού Επιτρόπου για τα θέματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια για τον εαυτό μου. Ποιος είμαι, ποια είναι η εμπειρία μου και γιατί πιστεύω ότι μπορείτε να μην εμπιστευτείτε. Τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής μου τα πέρασα σε ένα σοβιετικό γκουλάκ, σε ένα γκουλάκ του Στάλιν, στην Βόρεια Σιβηρία, στον Ακτικό Κύκλο. Γεννήθηκα εκεί μέσα σε μια οικογένεια εκτοπισμένων δημοσίων υπαλλήλων από τη Λιθουανία. Όπως ο πατέρας μου, από τα νιάτα μου έχω αγωνιστεί εναντίον της Σοβιετικής καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποστήριξα πάντα την αλήθεια, την δικαιοσύνη και την ισότητα. Δυο φορές συνελήφθη και ανακρίθηκα από την ΚΑΓΕΜΠΕ. Αγωνίστηκα για την ανεξαρτησία της Λιθουανίας και είμαι υπερήφανος που είμαι ένας από τις συντάκτες της δήλωσης για την ανεξαρτησία και το σύνταγμα της χώρας μου. Για μένα, ο αγώνας εναντίον του εξτρεμισμού και των ολοκληρωτικών καθεστώτων είναι κάτι το οποίο συνάδει με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανθρώπινες αξίες. Υποστηρίζω λοιπόν τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευμάρεια. Και η πολιτική μου φιλοσοφία είναι η σοσιαλδημοκρατία. Δεν έχουμε πρώτη φορά στις Φρυξέλλες. Ήμουν επικεφαλής αντιπροσωπείας της Λιθουανίας στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης υπό τον Ζισκάρ Δεστέν. Ο Τζούλιαν Αμάτο και ο Ζαν Λικτεάν ήταν αυτοί που με δίδαξαν πώς να καταλήγω σε συμβασμούς και συμφωνίες για την Ευρώπη. Γνωρίζω πάρα πολλούς από τους τωρινού ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λίγα λόγια στα λιθουανικά. Οι σπουδές μου ήταν στην ιατρική και είμαι καρδιοχειρουργός. Για 23 χρόνια η ζωή μου ήταν να σώζω ζωές. Ήθελα πάντα να δίνω στους ανθρώπους την ευκαιρία να έχουν μια πιο υγιεινή ζωή. Αυτό είναι το πάθος μου, αυτό είναι η αποστολή μου. Το Μάιο εφέτος εξελέγει αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας. Το άλλο μου πάθος είναι η ιστορία. Σπούδασα την, σπούδασα την ιστορία και έχω ζήσει στο πετσί μου ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας, από τα γκουλάκ μέχρι τον υποψήφιο επίτροπο. Αυτός είναι μεγάλος δρόμος για να διατρέξει κανείς σε μια σύντομη ζωή. Είμαι πολιτικός και νιώθω εμπιστοσύνη και υπερηφάνεια γιατί με εξέλεξαν έξι φορές οι συμπατριώτες μου στην περιοχή του Βίλνιους. Και υπήρξα αναπληρωτής ε, πρόεδρος της Λιθεωνικής Βούλης και Υπουργό Υγεία καθώς και Επικεφαλής Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι η υποψηφιότητά μου υποστηρίζεται από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο. Τώρα έρχομαι σε ορισμένε από τι προτεραιότητε, τι οποίε θα εστιάσω στα επόμενα πέντε χρόνια. Το να προωθήσουμε την οικονομική ανάκαμψη τη Ευρώπη είναι ένα κέριο στόχο και είμαι πεπισμένο ότι οι πολιτικέ στον τομέα τη υγεία και των τροφίμων, τη ασφάλεια των τροφίμων μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο εδώ. <clears throat> Α ξεκινήσω με το θέμα τη υγεία. Η υγεία είναι ένα βασικό στοιχείο τη κοινωνική οικονομία αγορά. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια νέα όθηση για την υγεία στην Ευρώπη γιατί οι δαπάνες για την υγεία δεν είναι μονάχα δαπάνες. Η έγκαιρη και η παγκόσμια οικουμενική πρόσβαση στην περίθαλψη είναι μια επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην παραγωγικότητα. Πρέπει να σκεφτούμε πέραν τη οικονομιστική άποψη των δαπανών. Πρέπει να δούμε τους ανθρώπους και την υγεία τους σαν ένα κύριο στοιχείο ενεργητικού για την κοινωνία μας. Γι' αυτό υποστηρίζω τη συνένωση των προσπαθειών των κρατών μελών για να έχουμε περισσότερες επενδύσεις στην υγεία και να σώσουμε ζωές. Μπορούμε από κοινού να κάνουμε περισσότερα, μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα και να βοηθήσουμε του πολίτε μα να ζήσουν πιο υγιεινές ζωέ. Θα συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη για να του βοηθήσω να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των υγειονομικών συστημάτων, ώστε με τον τρόπο αυτό να υπάρξει ισοδύνα, ισοδίκαια πρόσβαση στην ε, περίθαλψη για όλου του πολίτε. Για τον στόχο αυτό θέλω να δημιουργήσουμε και ένα σύστημα αξιολόγησης που να υποστηρίζει την παγκόσμια, την οικουμενική πρόσβαση στην υγεία, να ενισχύει την πρωτογενή περίθαλψη και να προωθεί την υγεία και την ασφάλεια. Αυτή είναι μερική από τους στόχους μου. Οι προτεραιότητες μου λοιπόν για τη δημόσια υγεία είναι πράγματι η προώθηση της ε, υγείας, η πρόληψη και η προστασία. Αλλά αυτό για όλους. Θέλω να ενισχύσω την προληπτική ιατρική. Όσο περισσότερο εστιάζουμε στα υγειονομικά μας συστήματα για την πρόληψη, τόσο λιγότερο θα κοστίσει η θεραπεία σε 10-20 χρόνια. Δεν είμαι εδώ για να σας πω να σταματήσετε το κάπνισμα ή να μην πίνετε. Απλώς θέλω να σας πω πόσο καλύτερη μπορεί να είναι η ζωή χωρίς να καπνίζει κανείς και χωρίς να κάνει κατάχρηση αλκοόλ. η προώθηση μιας υγιεινούς μορφής ζωής είναι μεγάλη σημασία. Αν μπορέσω να αποκομίσω την εμπιστοσύνη σας θα κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω τους πολίτες από υγειονομικές κρίσεις ή κρίσεις τροφίμων στο μέλλον. Θα εξασφαλίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη και μπορεί με μεγάλη ταχύτητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση που έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Η επιδημία της έμπολα είναι μια σαφής προειδοποίηση του κινδύνου που μπορεί να προκληθεί από τις λοιμώδεις ασθένειες και τις ανάγκες να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη της βοήθειάς μας. Πρέπει να βοηθήσουμε επίσης τους πολίτες μας να γεφυρώσουν το χάσμα υγείας στην Ευρώπη. Εγώ θέλω να υποστηρίξω τις αρχές της ισότητος και της αλληλεγγύης. Υγεία για όλους και όλοι στον σκοπό της επίτευξης καλύτερης υγείας. Τέλο, τέλος θέλω να υπάρξει μια πλήρης εφαρμογή των διαμεθοριακών οδηγιών για την υγειονομική περίθαλψη. Μπορείτε να βασιστείτε σε μένα να υποστηρίξω τα δικαιώματα των ασθενών. Θα παρακολουθήσω επίσης την εφαρμογή της οδηγίας για τα καπνικά προϊόντα και θα πάρω και τις απαραίτητες ε, για τους εφαρμοστικούς ε, νόμους. Συνεχίζω στα πολωνικά τώρα για την ασφάλεια τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια καλώς ανεπτυγμένη πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων. Πρέπει όμως να παραμείνουμε επάγρυπνοι και να αντιμετωπίσουμε <clears throat> τις ενδεχόμενες κρίσεις. Προτεραιότητά μου είναι να εξασφαλίσω ότι οι πολίτες της Ευρώπης θα έχουν τα πιο ασφαλή τρόφιμα στον κόσμο. Χρειαζόμαστε τα ασφαλή τρόφιμα ώστε να εξασφαλίσουμε και την υγεία των πολιτών μας. Τα πρότυπά μας για την ασφάλεια τροφίμων είναι επίσης θετικά για τους Ευρωπαίους παραγωγούς γιατί μας επιτρέπουν να είμαστε ανταγωνιστικοί στις παγκόσμιες αγορές. Θέλω λοιπόν να αξιολογήσω κατά πόσο μπορούμε να απλοποιήσουμε τους κανόνες μας σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων. Ο τομέας αυτός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μπορεί να συμβάλλει σε μεγαλύτερη ευμάρεια καθώς και σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αυτό ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά του τομέα παραγωγής τροφίμων. Περαιτέρω όμως πρέπει να δούμε και το θέμα των υγιεινών τροφών, γιατί είναι και ένας παράγων από τον οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η υγεία των πολιτών μας. Θα χρησιμοποιήσω κάθε ευκαιρία για να διατηρήσω και να βελτιώσω το σύστημα αυτό, εργαζόμενος με όλους τους εμπλεκομένους. Όλοι έχουν να διαδραματίσουν ένα ρόλο στο θέμα αυτό, από τους παραγωγούς τροφίμων μέχρι τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Και όλοι θα μπορέσουν να αποκομίσουν ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Μας έδειξε η πρόσφατη ιστορία ότι μπορεί να υποσκαφθεί η εμπιστοσύνη στα τρόφιμα από τις απάτες και τις κρίσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να μειώσουμε το περιθώριο για απάτες και θα υπάρχει ισότητα ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Μέσα στα πρώτα έξι, μέσα στους πρώτους έξι μήνες της εντολής μου θα ε, περάσω σε μία αναθεώρηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ακολουθώντας τη γραμμή που έχει χαράξει ο Ζαν Κλοντ Ιούγκερ. Επίσης, θα συνεχίσω τις ε, συζητήσεις που έχουν να κάνουν για την πρόταση περαιτέρω καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Επίσης, θα εξετάσω όλες τις προτάσεις που θα συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Θα ήθελα επίση να τονίσω ιδιαίτερα το πακέτο μέτρων που έχει να κάνει με την υγεία των ζώων, την ε, υγεία των φυτών και τους ε, φυτογειονομικούς ελέγχους που θα πρέπει να ενισχυθούν και συγχρόνως να απλοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο της καλύτερης ε, νομοθεσίας. Εάν εκλεγώ θα συνεχίσω αυτέ τι προσπάθειε με έναν τρόπο ο οποίο είναι διάφανος. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εταίρο μου στα θέματα αυτά. Είμαι έτοιμο να δώσω τι ε, επιλογέ που πρέπει να έχουν οι πολίτε μα εδώ και 50 χρόνια Αγωνίζομαι για αυτόν τον σκοπό και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Αν έχω την εμπιστοσύνη σα θα εργαστώ μαζί σα που είσαστε οι εκπρόσωποι των λαών τη Ευρώπη. Πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στου πολίτε μα και να επιτύχουμε μεγαλύτερη, καλύτερη υγεία ξέρουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ας το πράξουμε, ας προχωρήσουμε. Thank start... Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε με τον πρώτο κύριο ερωτήσεων μεγάλης διαρκείας. Πρώτος είναι ο Πίτερ Λίζη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε υποψήφιε Επιτροπέ, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Μιλήσατε για τις κοινέ αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα τον κλονισμό των ζώων, την κλωνοποίηση των ζώων. Γνωρίζετε πως ε, το Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένες απαιτήσει και ε, παρακολουθούμε επικριτικά την πρόταση της ε, Κομισιόν. Πώς τι σκοπεύετε να κάνετε για την κλωνοποίηση ζώων ε, για την διατροφή. Το δεύτερο είναι τι σκοπεύετε να κάνετε με τη μη εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος που αναφέρεται και στην Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βλέπουμε πως στον τομέα των κιτάρων και ιστών υπάρχουν δραματικές εξελίξεις, εμπόριο οαρίων ε, κτλ. Θα αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Επίτροπος. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τη δεύτερη ερώτησή σας που αφορά τα κύτταρα και τους Θα βασιστώ στη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων η οποία χάρτα δηλώνει σαφέστατα ότι τα ανθρώπινα σώμα και τα ανθρώπινα όργανα επουδενή δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου δεν μπορούν αντικείμενα ε, επιχειρηματικών συναλλαγών. Πιστεύω ότι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μας υποχρεώνει να σκεφτούμε τους τρόπους επίλυσης ε, των συγκεκριμένων προβλημάτων. Όσον αφορά την κλωνοποίηση ζώων για σκοπούς διατροφής και παραγωγή τροφίμων είναι περιπλοκότατο δεντολογικό ζήτημα και στο Κοινοβούλιο και στο ευρύτερο κοινό ακούμε ποικιλία απόψεων Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το τομέα όσον αφορά τις προτάσεις που έχουν τεθεί εν ίδια αντιδράσεως θα έλεγα ότι θα πρέπει προσεκτικά να επιδιωχθεί συμβιβαστική λύση γνωρίζω τη θέση του Κοινοβουλίου και γνωρίζω ποιες συζητήσεις αναμένουν. Please, Peter. Ε, σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την μη εμπορευματοποίηση του ανθρωπίνου σώματος, ε, ακούσαμε μια υπόσχεση. Όσον αφορά βεβαίως ε, την κλωνοποίηση, ε, υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο παρά τις διαφορετικές απόψεις ε, και η πλειοψηφία λέει πως δεν πηγαίνει αρκετά μακριά η πρόταση της Κομισιόν. Ως Επίτροπος λοιπόν θα φροντίσετε να υπάρξει μια αναθεώρηση αυτής της πρότασης της ε, Κομισιόν και να έρθετε κάπως πιο κοντά σε αυτά τα οποία προτείνει το Κοινοβούλιο. Η θέση μου είναι σαφέστατη. Είμαι ειλικρινής. Είμαι ειλικρινής ε, συζητητής, διαμεσολαβητής θα έλεγα. Προσπαθώ να συντονίσω τις διάφορες απόψεις θα πρέπει να καταλήξουν συμβιβασμούς που θα συγκεράζουν διαφορετικές απόψεις. Θα ήθελα να αναλύσω προσεκτικότατα τα προτινόμενα πακέτα και να προσπαθήσω να βρω την καλύτερη δυνατή λύση. Είμαι σίγουρος ότι η απόφαση θα ληφθεί συλλογικά, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συλλογικά κινείται και θα πρέπει να παρουσιάσουμε μια θέση η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα ο Ματίας Γκρότ για τους σοσιαλιστές έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Αντριουκάητης, μιλήσατε για πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Μια προτεραιότητα που θέλετε να έχετε ως ε, επίτροπος πρέπει να είναι κάτι αυτονόητο για όλους τους πολίτες της Ένωσης πώς θα βοηθήσετε τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες υγείας. Είπατε κάποια πράγματα. Και βεβαίως εδώ πέρα πρέπει να δούμε και τη διασυνοριακή υπαροχή υπηρεσιών υγείας. Και στην εφαρμογή. Υπάρχει η νομοθεσία, εγώ ζω σε μια μεθοριακή περιοχή, αλλά είναι δύσκολο ακόμα να εφαρμοστεί το πράγμα αυτό στην πράξη. Γιατί είναι πρόβλημα ακόμα η εφαρμογή. Και τι θα κάνετε ως Επίτροπος Υγείας για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα συγκεκριμένα. Εδώ ασχολούμαστε με ένα θέμα το οποίο απαιτεί μια απάντηση. Η απάντηση θα μας λέει του πότε θα πλησιάσει περισσότερο Ευρώπη τους πολίτες. Είναι κάτι σημαντικό αυτό για εκατομμύρια εκα... ανθρώπους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Η οδηγία υιοθετήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 2013 έπρεπε να σωματωθεί στις εθνικές ένομες τάξεις ήδη, πέρασε ένας χρόνος, πρέπει να δούμε τι συνέβη και αν χρειάζεται πρέπει να ξεκινήσουμε διαδικασίες κατά παράβαση. Δεν μπορούμε πλέον να ε, κολυσιεργούμε. Θα μπορούσα να σχολιάσω εκτενώς το θέμα, θα μπορούσα να πω ότι ε, τα εθνικά κέντρα διαβούλευσης έπρεπε να δημιουργηθούν, σημεία επαφής έπρεπε να αποφασιστούν, έπρεπε να θεσπιστούν συγκεκριμένα κριτήρια, να προετοιμαστούν πληροφορίες, θέματα που σχετιζόταν με διαδικασίες αποζημίωσης έπρεπε να επιληθούν, άρα είναι ευρύτατο ζήτημα. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκινήσουμε είναι σημαντικό το ζήτημα, θα μπορούσαμε να βρούμε πολλά σχετικά παραδείγματα στην Ισπανία, στη Λιθουανία, στην Ιρλανδία. Ε, κυρίως όσον αφορά ανθρώπους που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές. Πολύ συχνά μπορούν να τύχουν περίθαλψης 80 χιλιόμετρα εντός της άλλης χώρας. Σε άλλη περίπτωση στα 20 χιλιόμετρα σε διαφορετική χώρα. Πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση και γρήγορα. Αυτό είναι διαμφισβήτητο. Όσον αφορά την διασυνοριακή ε, απειλή, επιδημίες, πανδημίες κλπ. Ε, το όλο πακέτο είναι πάρα πολύ ευρύ και θα το επεξεργαστεί δεόντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ματίας, έχει συμπληρωματική ερώτηση, όχι, ευχαριστώ. Και τώρα για την ομάδα ECR θα δώσω το λόγο σε συνάδελφο Γκέρλινγκ. Ή θα μιλήσει πρώτα ο συνάδελφος Πιέκα. Γκέρλινγκ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα για τους υγειονομικούς ισχυρισμούς. Η, η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας είναι κάπως προβληματική κάποια τρόφιμα επηρεάζονται. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν στοιχεία για να υποστηρίξουν αυτούς τους ισχυρισμούς, αλλά οι μέθοδοι της Κομισιόν και της ΕΦΣΑ σημαίνουν πως δεν ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς. Βεβαίως χρειάζεται κάποια βελτίωση στην διαδικασία και μάλιστα η Κομισιόν το έχει πει πολλάκις ε, και ενώπιον της Επιτροπής μας και σε εμένα προσωπικά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ο Επίτροπος σκοπεύει να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους για να αναθεωρήσει αυτή τη διαδικασία όπως μας υποσχέθηκαν. Θα ξεκινήσει η αναθεώρηση σύμφωνα με το πρόγραμμα το 2015. Θα τηρήσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα και ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας για την αναθεώρηση αυτή. Ε, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. σαν υποψήφιος ε, επίτροπος δεν θα μπορούσα σε αυτή τη φάση να σας πω πόσα συγκεκριμένα ζητήματα καλύπτονται από τον κανονισμό. Χρειάζεται χρόνος για να καλυφθούν όλες οι λεπτομέρειες. Σαν γιατρός γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η μέτρα πρόληψης και προώθηση της υγείας, η προφύλαξη εν γέννη, όλα αυτά αποτελούν ακρογωνίο λίθο της προσπάθειας και δίνουν προστιθέμενη αξία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρμοδιότητες εθνικών κυβερνήσεων είναι πολύ ευρείες όσον αφορά την περίθαλψη του τομέα της υγείας και σε άλλους τομείς. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε αυτές τις αρμοδιότητες και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε ούτως ώστε οι αποφάσεις μας να δίνουν τη θέμενη αξία και οι εθνικές και οι ευρωπαϊκές αποφάσεις να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Βέβαια, είμαι υποχρεωμένος να ακούσω τις θέσεις των κρατών μελών, ε, να συζητώ και να συμβιβάζομαι. Είμαι γενικά ανοιχτός άνθρωπος και κάποιος που γνωρίζει εις βάθος αρκετούς τομείς, άλλους τομείς δεν τους γνωρίζω τόσο καλά. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τα κράτη-μέλη και να προσπαθήσω να, δω τι είδους αναθεώρηση χρειαζόμαστε, τι είδους μεταρρύθμιση θα πρέπει να κάνουμε να συζητήσουμε το θέμα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτως ώστε η διαδικασία να είναι πιο δημοκρατική και πιο ανοιχτή. Ε, όλοι θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες, εταίροι, ούτως ώστε να έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα υγείας και η πρόληψη να αποτελεί βασικό μας στόχο. Θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών στα πέντε χρόνια αν κινηθούμε ότι τρόπος. Κυρία Γκέρλινγκ, συμπληρωματική ερώτηση. Παραμένω στο ίδιο ερώτημα που έθεσα γιατί δεν πήρα πραγματικά απάντηση. Αυτό το οποίο ρώτησα ήταν το εξή. Υπάρχει αυτή η διαδικασία αναθεώρηση, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει το 2015. Ανεξάρτητα από το πώ θέλετε να συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη, αυτό είναι θέμα του Κοινοβουλίου. Εμεί εκπροσωπούμε του πολίτε. και είναι σημαντικό θέμα για μα αυτό ο κανονισμό. Θα, δει, θα τηρήσετε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα αυτό του 2015 ή όχι. Απάντηση. Η απάντησή μου είναι, είναι ανοιχτή και ειλικρινής. Πρέπει να παραμείνουμε στο χρονοδιάγραμμα αυτό, είναι σίγουρο. Πρέπει να συζητήσουμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά τώρα δεν είμαι σε θέση να σας πω ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερε πολυπλοκότητε. Είμαι έτοιμο όμω, να συζητήσω όλα αυτά τα θέματα με το Κοινοβούλιο μέσα στο χρονοδιάγραμμα αυτό. Και μέσα στην αναθεώρηση θα πρέπει να πάρουμε συλλογικέ αποφάσεις για τα θέματα αυτά. Και τώρα για την Άλτε, Φρέντερικ Ρίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι κύριε Επίτροπε, <clears throat> υποψήφια Επίτροπε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το τελευταίο ευρωβαρόμετρο από το 2010 βέβαια είναι κάπως ε, πεπαλαιωμένο, πρέπει να το επικαιροποιήσουμε. Όλα τα στοιχεία έχουν την ίδια τάση. Μόνο 21% λέει το ευρωβαρόμετρο των Ευρωπαίων θεωρούν ότι είναι ασφαλή τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα για την υγεία μας και για τις ε, μελλοντικέ γενιές. Οι απαντήσεις που δώσατε ήταν σαφείς. Ο κύριος Ιούγκερ ζήτησε να αναλάβετε δράση μέσα στους επόμενους έξι μήνες και ήταν σαφείς και σε αυτά που είπε και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο και ενώπιον των πολιτικών ομάδων. Έδωσε ένα σαφές μήνυμα ότι η πολιτική του φιλοδοξία είναι να κινηθεί προ την κατεύθυνση αυτή. Θα τώρα να δω πώ εσεί θέλετε να υλοποιήσετε αυτή την πολιτική δέσμευση για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού που είναι κομμάτι τη εντολή σα, ποιε μεθόδου θέλετε να χρησιμοποιήσετε και έχετε απαντήσει μέχρι τώρα για... σε γενικό επίπεδο θα ήθελα να σας όμως πιο συγκεκριμένος στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Κάιτης εγώ περίμενα κάποιος να μου θέσει αυτό το ερώτημα γιατί την τμήμα της εντολής που έχω αναλάβει από τον πρόεδρο Γιούνκερ και αν η νέα Κομισιόν μπορεί να ξεκινήσει το έργο της πράγματι την 1η Νοεμβρίου, από την πρώτη στιγμή εγώ θα πρέπει να αναλάβω μέτρα και να εξετάσω όλο το πακέτο νομοθετημάτων που έχουν να κάνουν με αυτή τη διαμάχη σε σχέση με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η Κομισιόν δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση η οποία παραγνωρίζει τις θέσεις των κρατών μελών. Νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την επικουρικότητα που έχουν τα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά και οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί από την Κομισιόν θα πρέπει να περιλαμβάνεται μέσα στην εντολή που έχει να κάνει με την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη χωρίς όμως να έλθουν σε σύγκρουση με τα κράτη-μέλη. Για τις λεπτομέρειες θα πρέπει να σχεδιάσουμε όλο αυτό το έργο εγκαίρως και ο στόχος μου είναι από τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλέκεται πλήρως ώστε να έχουμε ένα κοινό σχέδιο δράσης. Μίλησατε για κάποια κάτι μέλη τα οποία ε, αντιτίθενται σε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι λίγα κράτη-μέλη, είναι 19 τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν κρατήσει αντίθετη θέση για την έγκριση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Όποια και να είναι η θέση μας, υπάρχει μια κατάσταση αυτή τη στιγμή εμπλοκής. Δεν υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσει. Και ένα άλλο ερώτημα, πιο εικονοκλαστικό αν θέλετε. Τα θέματα αυτά των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, μήπω θα ήταν καλύτερο να τα αντιμετωπίσουμε σε εθνικό και ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί υπάρχουν διαφορετικέ κουλτούρε σε σχέση με τα θέματα αυτά στι χώρε μα και τι περιοχέ μα. Απάντηση. Ναι, κατανόησα την ουσία της ε, ερωτήσεώς σας. Σίγουρα η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ευρώπη αποτελεί τεράστιο φιλοσοφικό ζήτημα. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος βιοπικιλότητας. Βλέπουμε διαφορές ε, που υπάρχουν μεταξύ περιοχών και αν θέλουμε να παρέμβουμε σε αυτήν την τεράστια βιολογική ποικιλομορφία και την αρμονία και αν αλλάξουμε τις ισορροπίες, αυτό θα είναι κάτι επιβλαβές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι σοβαρό ζήτημα. Τώρα αν μιλήσουμε για συγκεκριμένα πρακτικά βήματα, όταν είναι σαφής η θέση των κρατών μελών, πράγματι αλήθεια είναι ότι αποφάσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και υπάρχουν και διασυνοριακά ζητήματα βέβαια διότι όλοι έχουμε σχέση μεταξύ μας αλλά πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ και τώρα για την ΚΟΕ η συνάδελφος Κονέτσνα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε Επίτροπε. Στην επιστολή σας, στις γραπτές απαντήσεις, σωστά αναφέρεται πως έχουμε πολύ αυστηρές προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των τροφίμων και ταυτόχρονα λέτε πως είναι προτεραιότητά σας να διατηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές. Από την άλλη, θα ε, υιοθετήσουμε προσεχώς την συμφωνία TTIP, την ε, Διατλαντική, που έχει ακόμα πολλά ανοιχτά ζητήματα και εγώ θεωρώ πως είναι μια συμφωνία που εγκυμονεί κινδύνους ε, για την υγεία και την ζωή των πολιτών στην Ευρώπη. Πώς θα αποτρέψετε ως Επίτροπος το να κινδυνεύσουν αυτές ακριβώς οι υψηλές προδιαγραφές ε, της περίθαλψης ε, της ιατροφαρμακευτικής των ε, Ευρωπαίων ασθενών. Ευχαριστώ. Ως γιατρός αντιλαμβάνεστε πως η απάντησή μου είναι όχι σε οποιαδήποτε εξασθένηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών είτε μιλάμε για την ασφάλεια των τροφίμων, είτε για την υγεία. Ήταν σαφής η θέση επίσης ε, του Προέδρου της Κομισιόν, ο οποίος είπε ότι δεν θα θυσιάσει ποτέ την ασφάλεια των τροφίμων ή την υγεία για χάρη του ελευθερου Νομίζω ήταν σαφές το μήνυμα. Προσωπικά δεν μπορώ να κάνω κανέναν συμβιβασμό τέτοιου είδους. Είτε μιλάμε για τις ορμόνες στο κρέας, είτε για τα χλωριωμένα κοτόπουλα. Η απάντηση είναι η ίδια. Ε, οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ψηλότερες και το καλύτερο παράδειγμα του πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία του κόσμου σε μια εποχή βιομηχανοποιημένη. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και εγώ τι σημειώνω αυτή την υπόσχεσή σας. Από την άλλη βεβαίως δεν θα είναι εύκολη υπόθεση και έχω άλλη μία ερώτηση ε, που επίσης αφορά την ασφάλεια. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε διάφορα είδη τροφίμων, διαφόρων ειδών. Μιλάω κυρίως για την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Τι θα κάνετε για τις εταιρείες εκείνες οι οποίες σε διαφορετικές αγορές ε, πουλάνε διαφορετικά προϊόντα με διαφορετικά συστατικά. Ευχαριστώ. Πρέπει να πω πως ε, η εποπτεία της ποιότητας ε, των ε, τροφίμων γίνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για εσωτερική αγορά, κοινέ προδιαγραφές και για την υποχρέωση τήρησης αυτών των προδιαγραφών είτε είμαστε στην Πολωνία, Λιθουανία είτε στην Πορτογαλία. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα ελέγχου. Αντιλαμβάνομαι το ζήτημα το οποίο αναφέρεται για τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και τα τρόφιμα και όλα τα σχετικά ζητήματα και πράγματι πρέπει να παρακολουθούμε το ζήτημα. Καμιά φορά συμβαίνει να μην ε, είναι ακριβώ οι ίδιες οι προδιαγραφές ε, και να παίζουν κάπου με τις οριακές τιμές, αλλά θα είμαι πολύ δραστήριος στον τομέα αυτό, σας το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους ε, συνάδελφους Στάες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Θα συνεχίσω και εγώ με το θέμα της TTIP, της συμφωνίας αυτής με τη ΣΥΠΑ. Εγώ θα σημειώσω την υπόσχεσή σας ότι δεν θα συμβιβαστείτε καθόλου στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και ο καθένας αντιλαμβάνεται πως η Κομισιόν δεν πρόκειται να αποσύρει ξαφνικά την ε, οδηγία για τις ορμόνες ή τις γενετικά τροποποιημένους ε, οργανισμούς. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και η μελλοντική νομοθεσία. Και βλέπουμε εδώ πέρα πως η προηγούμενη επιτροπή, η επιτροπή Μπαρόζο, έφερε κάποιες προτάσεις ε, για τη χλωρίωση, για τον κλονισμό, για το γαλακτικό οξύ και το τι θα γίνει με τα κλωνοποιημένα ζώα ε, και είχαμε ακριβώς πίεση λόγω των διαπραγματεύσεων του ελευθέρου εμπορίου. Η ερώτησή μου είναι σαφής, τι θα κάνετε για να ε, επιτύχετε αυτούς τους στόχους και να αντισταθείτε σε αυτή την πίεση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να κάνω το εξή σαφέ σε όλους. Η διαφάνεια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να είναι απόλυτα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η διαφάνεια αυτή και θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις και κλεισμένων των θυρών. Θα πρέπει να έχουμε σαφήνεια τι είναι το αντικείμενο σε διαπραγμάτευση σε κάθε χώρο και επίσης αυτό θα πρέπει να περάσει και να υποβληθεί στα Εθνικά Κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τέλος. Όταν φτάσει η διαδικασία αυτή, φυσικά υπάρχει ανάγκη κύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα να εμπλακεί, να εμπλακούν οι επιτροπές και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσετε εσείς σαν Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Γεωργίας. Αλλά δεν μπορούν αυτές οι επιτροπές να βγουν από τη διαδικασία. Εγώ είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Όπως ξέρετε είμαι ιατρός, έχω, ε, έχω δώσει τον υποκρατικό όρκο και για όλους αυτούς τους λόγους Τονίζω ότι δεν πρέπει να υπονομευθεί το επίπεδο προτύπων των ε, τροφίμων μας και των προϊόντων μας και ξέρω ακριβώς που θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επάγρυπνοι για τα θέματα αυτά. Ε, ε, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ερώτημα του κυρίου Λίζε μαζί με τον κύριο Λίζε και άλλου συναδέλφου. παρακολουθήσαμε την τελευταία αποφάση τη διαπραγμάτευση για το καινοτόμα τρόφιμα που διακόπηκε το Μάρτιο του 2012 ακριβώς στο ζήτημα του τι θα κάνουμε με το κρέας κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους. Και το Κοινοβούλιο είπε πως θέλουμε ξεκάθαρη σήμανση και προτάσεις της Κομισιόν. Στο τέλος προηγούμενου έτους έφερε προτάσεις η Κομισιόν και προς έκπληξή μας διαπιστώσαμε πως δεν αναφέρεται τίποτα για σήμανση και ακόμη χειρότερα σε ένα από τους δύο φακέλους η νομική βάση είναι τέτοια που δεν επιτρέπει ρόλο του Κοινοβουλίου στην συναπόφαση. Είπατε στον κύριο Λίζε πως ε, θα διευκολύνετε την κατάσταση, θα είστε διαμεσολαβητής, θα βρείτε έναν συμβιβασμό. Κύριε Υποψήφιε Επιτροπέ, καλύτερο είναι νομίζω αυτή τη στιγμή μαζί με τη νέα Κομισιό να αποσύρετε αυτή την πρόταση και να φέρετε μια καινούρια για το κρέας κλωνοποιημένων ζώων για να ξεκινήσουμε από μια καινούρια βάση. Για το θέμα αυτό και πάλι μπορώ να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν μπορώ βέβαια να προκαταλάβω τι θα προκύψει στο τέλος της διαδικασίας αυτής. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το τι θα κάνουμε για τον τομέα αυτό. Εδώ τίθεται ένα θέμα δεοντολογίας, ένα θέμα ηθικής το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Και από βιολογική άποψη είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ πολύπλοκο. Η, η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός της δεύτερης και της τρίτης γενιάς και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις για τα θέματα αυτά και θα προσπαθήσω να βρω μια, ένα κοινό έδαφος. Ξέρω πόσο μεγάλη ευθύνη φέρω για το θέμα αυτό και θα συνεχίσω τις προσπάθειές μου προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ για την EFTT, ε συνάδελφος Ματζουρόνης έχει το λόγο. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, υποψήφιο επίτροπε, καταρχάς σας καλωσορίζω εδώ, σας εύχομαι καλή επιτυχία για το επόμενο βήμα που θέλετε να κάνετε. Σαν πρώην υπουργό Υγείας, ξεκινήσατε πολλές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ε, υγείας. Κυρίως όσον αφορά την προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας στην Λιθουανία. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, συνεπώς. Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η φυγή εγκεφάλων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σαν πρόβλημα, κυρίως στον τομέα της υγείας. Όταν οικονομικά πιο αδύναμες χώρες ετοιμάζουν ειδικού με χρήματα του προπολογισμού του και οι επιστήμονε μετά φεύγουν για πλουσιότερε χώρε. Και διαμορφώνεται η εξή κατάσταση. Οι φτωχότερε χώρε έχουν χειρότερη πρόσβαση όσον αφορά την ε, περίθαλψη. Το ίδιο ισχύει και στην Λιθουανία, θα το γνωρίζετε. Ε, καταλαβαίνω πολύ καλά το δικαίωμα της ελεύθερης ε, διακίνησης, όμως το αναγνωρίζετε το πρόβλημα της φυγής εγκεφάλων στον τομέα της υγείας και τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ε, Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, το πρόβλημα πράγματι της διαρροής ε, κεφάλων όπως λέμε είναι πραγματικό. Σχετίζεται βεβαίως με τις διαφορές στους μισθούς, στις ευκαιρίες σταδιοδρομίας ε, και ε, στις, στην οικονομία. Οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες πράγματι εκπαιδεύουν με δημόσιο χρήμα ειδικού ε, επενδύουν δηλαδή στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μετά φεύγουν και αφήνουν τις χώρες σε μια χειρότερη κατάσταση. Τα ζητήματα λοιπόν του κοινωνικού ντάμπινγκ είναι πάρα πολύ επίκαιρα και σε άλλα επαγγέλματα. Νοσηλευτές παραδείγματος χάρη. Στη χώρα μου, στη χώρα την οποία γνωρίζω καλύτερα, εμείς εκπαιδεύουμε πολλούς νοσηλευτές ε, και δεν έχουμε αρκετές ε, γιατί φεύγουν. Το ίδιο και με τους γιατρούς. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τον ε, προγραμματισμό της αγοράς εργασίας και να βασιστούμε βεβαίως και στην κοινωνική χαρτά. Όλα αυτά έχουν σχέση με την εντολή μου. Νομίζω πως ε, είναι αρμοδιότητα άλλων επιτρόπων, των αρμοδίων για την εκπαίδευση, της κοινωνικές πολιτικές. Νομίζω πως ε, πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά αυτό το θέμα. Σας... Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συμπληρώσω την ερώτησή μου Δηλαδή πώς να το εκλάβω αυτό που είπατε, ότι υπόσχεστε εδώ και τώρα να συνεργαστείτε με άλλους επιτρόπους στον τομέα αυτών Και ότι εσείς ο ίδιος θα ξεκινήσετε την προσπάθεια εξέβρεσης λύσεων. Θα μπορούσατε να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη για το εξή θέμα. Όταν υπάρχουν κοινωνικά χάσματα, Και όταν πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές που υπάρχουν στον τομέα αυτό. Άμα θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους να έχουν κάποια προοπτική για το μέλλον τους, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το θέμα χωρίς να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένοι από την Ευρώπη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη των πολιτών ε, στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εγώ σας έχω υποσχεθεί στον τομέα αυτό να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου και εδώ είναι ένα θέμα που δεν έχει να κάνει μοναχά με την ε, αποτελεσματικότητα του υγειονομικού συστήματος αλλά και για το μέλλον το οποίο θα δημιουργηθεί. Και θα για αυτά. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε τον πρώτο γύρο που πλευρά των συντονιστών, μάλλον των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο με τις ερωτήσεις των συναδέλφων της Επιτροπής Περιβάλλοντος να δώσω αμέσως το λόγο για αυτές τις σύντομες ερωτήσεις με μία απάντηση στη συνάδελφο Μπέτ Κόστιγκερ. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου αφορά την πρόταση κανονισμού για την εμπορία σπόρων. Μας είπατε πως μετά την εξέταση της θέσης του Κοινοβουλίου θα δείτε ποιος θα είναι ο καλύτερος ε, Δρόμο σου πρέπει να ακολουθήσετε. Πολύ ευγενικό αυτό. Είναι σαφής η θέση του Κοινοβουλίου. 650 βουλευτές απέρριψαν την πρόταση της Κομισιόν. Η Γεωργία χρειάζεται ανεξαρτησία στο θέμα των ε, σπόρων και βεβαίως να προστατευτεί η γενετική ποικιλομορφία. Γνωρίζετε πως το Κοινοβούλιο έχει μεγάλα προβλήματα με την γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν ε, οι μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι τι σκοπεύετε να κάνετε εδώ πέρα για να αντιμετωπίσετε τις αμφιβολίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αν θα μπορέσετε να φέρετε πραγματικά μια πρόταση η οποία θα ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία απαιτούνται στην πράξη. Σας ευχαριστώ. Το ζήτημα αυτό σχετίζεται με τη βιολογική ποικιλότητα. Στην χώρα μου έχουμε πράγματι προβλήματα καθώς οι τοπικές ποικιλίε παραμερίζονται και βλέπουμε πως υποβαθμίζεται η βιοπικιλότητα. Εντάξει, οι μικρές επιχειρήσεις δουλεύουν με τις ντόπιε ποικιλίε και είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν με τις μεγάλες. Γι' αυτό πιστεύω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί ακριβώς να προστατεύσει τα συμφέροντα των μικρών παραγωγών και αγροτών. Αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ τώρα να αναφέρω τη θέση του Συμβουλίου γιατί βεβαίως θα υπάρξει συζήτηση μεταξύ των δύο νομοθετών. Αλλά είμαι σίγουρος πως θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά προσεκτικά υπόψη έχοντας πάντα κατά νου πώς πρέπει να υπερασπιστούμε τις ε, τοπικές ποικιλίε. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρος Σάρμπου έχει το λόγο. Η Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι χρειάζονται κατεπηγόντως μέτρα όσον αφορά την παχυσαρκία των παιδιών θα ήθελα να ξέρω, έχετε συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Απευθυνόμαστε και προς άτομα με χαμηλότερο εισόδημα. Πώς θα προσεγγίσετε την ιδέα ανισότητας μεταξύ των συστημάτων υγείας που υπάρχει στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν πολύ ωραίο θα μπορούσα να σας δείξω μια εικόνα στις οθόνες. Πώς αντιδρά ένα παιδί τριών ετών σε σχέση με ένα προϊόν που βλέπει στην ε, τηλεόραση να διαφημίζεται παραδείγματος χάρη και πώς, μπορεί να προκύψει ένας κίνδυνος για την ε, υγεία των παιδιών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα σήμερα. Βλέπουμε ότι αυξάνεται ο αριθμός των παχύσαρκων παιδιών και αν συνεχίσει αυτή η τάση, σε 30 χρόνια θα είμαστε σε μια κατάσταση πανδημία σε σχέση με την παχυσαρκία. Ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάποιες μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Θα είναι πιο σοβαρό πρόβλημα και από τις λοιμώδεις ασθένειες και τον καρκίνο η παχυσαρκία αυτή. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες για το θέμα αυτό και εγώ ως ιατρός γνωρίζω τι σημαίνει αυτό για την υγεία των πολιτών. Χρειαζόμαστε κοινωνικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιείται η διαφήμιση. Πρέπει να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και με τους παραγωγούς τροφίμων και αυτούς που τα παρουσιάζουν και τα διαφημίζουν. Πρέπει να έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος για τα θέματα αυτά. Να υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση στα σχολεία για τους κινδύνους αυτούς. Πρέπει να αναλυφθούν λοιπόν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσουμε και την κοινωνική πτυχή του θέματος αυτού. Βλέπουμε ότι τα άτομα τα οποία έχουν χαμηλότερη μόρφωση έχουν μεγαλύτερη τάση να έχουν κακή διατροφή και να έχουν αρνητικές συνήθειες σε σχέση με την υγεία και έτσι δημιουργείται αυτό το χάσμα το κοινωνικό το οποίο ανέφερα προηγουμένως που μπορεί να γίνει μια επιδημία. Ευχαριστώ, συνάδελφε Πιάκα, για το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Υποψήφιε Επίτροπε. Δεχτήκατε την πρόταση να είσαστε υποψήφιος επίτροπος. Πρόταση που σας έκανε ο κύριος Γιούνκερ. Ο κύριος Γιούνκερ αναστάτωσε κάπως την όλη δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, χρειάζεστε κάποια εργαλεία για να εκτελέσετε τα καθήκοντά σας. Παραδείγματο χάρη και για να, κάνε, να εφαρμόσετε σωστή εποπτεία όσον αφορά ε, την Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Υγείας. Δυστυχώς, ο κύριος Γιούγκερ έδωσε την εποπτεία του φορέα αυτού στον Επίτροπο τον Αρμόδιο για θέματα βιομηχανίας. Και έτσι τίνω να πιστεύω ότι δεν υπερασπίζεται σωστά τα δικαιώματα των ασθενών. αλλά περισσότερο τις ε, φαρμακευτικές βιομηχανίες όσον αφορά τον έλεγχο της ΕΜΕΑ. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, διότι εσείς πρέπει να υπερασπίζεστε τα δικαιώματα των ασθενών και όχι των μεγάλων εκπροσώπων της ε, φαρμακοβιομηχανίας. Απάντηση. Η πρακτική μου, η εμπειρία μου που σωρεύτηκαν μετά τη συζήτηση για την, ε, για την συζήτηση για τα διάφορα φάρμακα, τα γενώσιμα κλπ. Και, και διαπιστώνοντα ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη αυτή η εμπειρία που συσσόρευσα είναι μεγάλη. Είχα πολλές επαφές με μεγάλες εταιρείες της φαρμακοβιομηχανίας και Πρέπει να συζητήσουμε την όλη κατάσταση. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερο σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων. Πρέπει να συζητήσουμε και με τη βιομηχανία το θέμα αυτό, διότι ασκούνται μεγάλες πιέσεις του προπολογισμού των κρατών μελών και αυτό το βλέπει ο καθένας. Είναι φανερό ότι οι συζητήσεις όσον αφορά τα συμφέροντα και τις διάφορες επιρροές πρέπει να είναι διαφανείς. Στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων και στις διάφορες υπηρεσίες του φορέα αυτού ε, έχουμε συζητήσει το θέμα και με την κυρία Μπιανκόσκα θα καταλήγουμε σε αποφάσεις από κοινού. Μια απόφαση μπορεί να θετηθεί μόνο όταν δύο επίτροποι υπογράψουν η πρόσβαση στα φθηνά φάρμακα και στα καινοτόμα φάρμακα για τους Ευρωπαίους είναι πολύ καυτό θέμα αυτές τις ημέρες και η δική μου εμπειρία μου λέγει ότι όλα ε, συνδέονται με την ε, αντίσταση των συστημάτων υγείας. Η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα επηρεάζεται από αυτό. Θέλουμε να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση για να βελτιωθεί και η ζωή των ανθρώπων. Νομίζω ότι θα βρούμε τελικά μια συμβιβαστική λύση με την κυρία Μπιανκόφσκα. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπέρντερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Η μείωση των ισοτήτων τη υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ύψιστη προτεραιότητα για τη στρατηγική και τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Κυρίω αντικατοπτρίζεται στο πακέτο για τι κοινωνικέ επενδύσει και το τρίτο πρόγραμμα για την δράση τη Ένωση στον τομέα τη υγεία μέχρι το 2020. Θα είσαστε υπεύθυνο γι' αυτό. Λοιπόν, και στο τομάτι αυτό για τι στρατηγικές δημόσια υγεία ε, στην εθνικό επίπεδο είναι και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και η υγεία θα πρέπει να βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού. Όμω, βλέποντα όλη την Ένωση, βλέπουμε ότι οι δείκτε όσον αφορά την υγεία δείχνουν τεράστιε διαφορέ και ανισότητε που επηρεάζουν του πολίτε. Δείχνουν σημαντικέ διαφορέ όσον αφορά την μητρική θνησιμότητα ε, των σεξουαλικά μεταδεδομένων ασθενειών και εμολύνσεων και πρόσβαση όσον αφορά ε, την περίθαλψη από πλευρά μεών. Λοιπόν, τι θα κάνετε όσον αφορά τα δικαιώματα της αναπαραγωγικής υγείας στο μελλοντική στρατηγική της Ευρώπης για την υγεία. Θα εξασφαλίσετε ότι τα εργαλεία και τα προγράμματα θα εφαρμόζονται σωστά. Δεσμεύεστε να υποστηρίξετε ε, μια προσέγγιση ευρωπαϊκή και ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τη σεξουαλική αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα όσον να υπάρχει ε, πρόσβαση στις πληροφορίες, στην πρόληψη κλπ. Και ε, ούτως να οδηγηθούμε σε μια μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών της Ένωσης. Κοιτάξτε. Εγώ πιστεύω ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη. Όχι μόνο γιατί είναι με στο χαρτοφυλάκιο ενός αντιπροέδρου. Υπάρχει πάντα κάποιος ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή όλων αυτών που συνάπτονται με τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Φυσικά <clears throat> και εγώ ως Επίτροπος για τα θέματα υγείας έχω μεγάλες ευθύνε για το θέμα αυτό και είμαι αρμόδιος για να το αντιμετωπίσω μαζί με τον αρμόδιο αντιπρόεδρο. Αυτό είναι ένα εγκάρσιο θέμα. Η προστασία λοιπόν των ασθενών και των δικαιωμάτων των ασθενών είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της, των προτεραιοτήτων της Κομισιόν. Αλλά είναι και η δική μου η εμπειρία ότι και εδώ θα πρέπει να μπορέσουμε να ακούσουμε και την άποψη των ασθενών για το ποια είναι η καλύτερη μεταχείριση και η θεραπεία που θα πρέπει, τις οποίες πρέπει να την χάνουν. Θα πρέπει λοιπόν με, να συζητήσουμε αυτό το θέμα της ικανότητας να επιλέγουν οι ίδιοι οι ασθενείς και όχι μόνο να παίζουν ένα ρόλο παθητικό, να συμμετέχουν στις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη θεραπεία τους και την υγεία τους. Και Νομίζω ότι είναι σαφές ότι είναι απαραίτητο σε κοινωνικό επίπεδο να λαμβάνονται ε, αποφάσεις αυτού του είδους και αυτό φάνηκε και στην έκθεση του Μάικελ Μάμοντ από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Ήταν σαφές σε παγκόσμιο επίπεδο πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός ρόλος για την διαμόρφωση της υγείας όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν τα επόμενα πέντε χρόνια να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία θα είναι και πολύπλοκα για να ξεπεράσουμε αυτό το κοινωνικό χάσμα που υπάρχει και θα πρέπει να μα φέρει αυτό και πιο κοντά στους πολίτες. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπόιλαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως γιατρό φαντάζομαι πως αντιλαμβάνεστε την ε, σημασία του ε, να βασίζεται η πολιτική σε επιστημονικά στοιχεία. Και βεβαίως εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας των Φίλων παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ε, ντομοκτώνα κτλ. Αλλά εδώ πέρα υποβαθμίζεται ο ρόλος της από συγκρόμενα συμφέροντα και σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, 41% όσων ερωτήθηκαν δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία των επιστημόνων λόγω της δουλειά που κάνουν για λογαριασμό του κλάδου. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πώς θα βελτιώσετε την ανεξαρτησία των δομών της υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων. Κοιτάξτε, στην καθημερινή μου ζωή εγώ συνάντησα ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, τον εμβολιασμό των παιδιών. Η παραγωγή των εμβολίων οι μελέτες, οι σχετικές και η έλλειψη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα των μελετών γιατί θεωρεί ο κόσμος πως ε, τις χρηματοδοτούν οι φαρμακευτικές εταιρείες και άρα δεν εμπιστεύονται τα αποτελέσματα. Είναι σοβαρό πρόβλημα αυτό και πρέπει να υπάρξει διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχουν ή δηλώσεις διαφάνειας, το ίδιο και για τις δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων. Η υπηρεσία θα μπορεί νομίζω να δίνει, να αιτιολογεί το γιατί απορρίπτονται κάποια πράγματα ενώ άλλα όχι και να είναι σαφές αυτό γιατί βεβαίως εύκολα χάνεται η εμπιστοσύνη και δύσκολα κερδίζεται. Και εδώ πέρα πρέπει να σκεφτούμε ένα σύνολο μέτρων και εργαλείων και το σημαντικότερο νομίζω είναι όταν αξιολογούνται επιστημονικά άρθρα να βασιζόμαστε σε σαφείς αρχές που θα είναι γνωστές στην κοινωνία, στους πολίτες, στο κοινοβούλιο. Πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η εμπιστοσύνη στις ε, αρχές, αλλιώς θα έχουμε διατροφικές κρίσεις και τέτοια πράγματα αυτή η δυσπιστία απέναντι στους επιστήμονες ε, υπάρχει σε διάφορους τομείς. Υπάρχει ένα ανεξάρτητο μέσο αξιολόγησης των μελετών, αλλά δεν επίθεται ο κόσμος και είναι τεράστιο το πρόβλημα. εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να, υπάρξει, να υπάρξουν αυστηρότερες προδιαγραφές. Σας ευχαριστώ. Άουκεν. Ευχαριστώ. Μου άρεσε η απάντησή σας για τη φαρμακοβιομηχανία, αλλά οι συντονιστές ανησυχούν για αυτό το ζήτημα. Και πώς ε, θεωρείτε ότι θα έχετε έλεγχο χωρίς ε, κάποια διοίκηση. Το άλλο, η άλλη ερώτησή μου αφορά τις ουσίες εκείνες οι οποίες ε, διαταράσσουν το ενδοκρινικό ε, και κάτι πρέπει να γίνει ε, για να ληφθούν μέτρα για αυτές τις ουσίες. Το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον σας δίνει σαφή έντολη και η ερώτησή μου είναι η εξής. Θα καταρτήσετε οριζόντια επιστημονικά κριτήρια κινδύνου για να αναγνωριστούν αυτές οι ουσίες ή όπως φοβόμαστε θα ε, έχετε μια πολιτική προσέγγιση για να μην επηρεαστούν οι επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, μιλήσατε για φόβο κτλ εμένα με συνέλαβε η KGB. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Σπούδασα ιατρική και το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μην ε, βλάπτουμε. Έτσι, είναι αυτά στον όρκο του Ιπποκράτη οι ουσίες αυτές που διαταράσσουν το ενδοκρινικό είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει να προσέξουμε, μην καταλήξουμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια ενδιάμεσα κριτήρια, ήταν η πρώτη που είχε τέτοια, ε, αλλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε βασισμένοι ε, σε επιστημονικά στοιχεία για να καταλήξουμε σε κάποια οριστικά κριτήρια. Είναι ευαίσθητος ο τομέας γιατί βεβαίως επηρεάζονται εδώ πέρα οι μελλοντικέ γενιές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αποφασισμένοι και να βασιζόμαστε σε αντικειμενικά κριτήρια. Έχουμε, όπως είπα, κάποια ενδιάμεσα κριτήρια και θα προσπαθήσω και εγώ να κινήσω τις διαδικασίες. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Πιεντετσίνη. Εδώ είμαι. Εκτιμήσαμε τη θέση σας κατά της διαφθοράς στον τομέα της υγείας και πάνω σε αυτό θέλουμε να επιθυμίσουμε σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ούτε στα νοσοκομεία. Επί πολιτική βάση διορίζονται οι γιατροί στα νοσοκομεία και όχι ε, με βάση τα προσόντα. Αυτό έχει αρνητικότατε συνέπειε όσον αφορά την υγεία των ασθενών και την παροχή των υπηρεσιών στο κόστο των συσκευών και των φαρμάκων. Και πολύ συχνά αυξάνονται δυσανάλογα όσον αφορά ε, ε, την περιπλοκότητα τομέα. Είπατε κάτι. Τι θέλετε να κάνετε για να υπάρχουν μια όμορφα ε, κριτήρια για την τιμολόγηση των φαραμάκων στα κράτη-μέλη και μεταξύ κρατών μελών και πώς θα γίνετε πώς θα αντιταχθείτε στη διαφθορά και στην πολιτική επιρροή στον τομέα της ε, υγείας. Patirtis, kurią tenka atsiremti, šitoj srity, aišku, ji gali būti Στον τομέα αυτό, Μπορεί να έχει συμβεί αυτό το οποίο είπατε, αλλά αυτό είναι θέμα το οποίο είναι θέμα αρμοδιοτήτων εθνικών. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει ότι σε όλους τους τομείς που έχουν να κάνουν με τον τομέα της υγείας και την αλυσίδα περίθαλψης να <clears throat> εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής αντιμετώπιση της διαφθοράς. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση. Δεν μπορούμε να έχουμε μεμονωμένες μονάχα ενέργειες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν και με τις δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον τρόπο αυτό. Ό,τι έχει να κάνει με αγορά φαρμάκων και εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται προς το συμφέρον το δημόσιο. <clears throat> θα πρέπει να ακολουθούν ένα κώδικα δεοντολογίας ο οποίος περιλαμβάνει την απόλυτη διαδικασία διαφάνειας. Και να εξασφαλιστεί ότι και η παράδοση και η προμήθεια των φαρμάκων στα νοσοκομεία θα πρέπει να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες. Εμείς μπορούμε φυσικά μονάχα να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη και να επιστήσουμε την προσοχή τους για το θέμα αυτό, γιατί παραμένει στην αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Και μπορούμε να ανταλλάξουμε και εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα αυτά. Στα προηγούμενα καθήκοντά μου εγώ είχα προωθήσει ιδιαίτερα την προσπάθεια αυτή. Όλα αυτά λοιπόν που λέτε για τις δημόσιες προμήθειες και την εφαρμογή αυτής της αρχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι φυσικά ένα θετικό βήμα, αλλά φυσικά πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ήδη κάνει μια συμφωνία για το λεγόμενο pooling και sharing των ε, ε, εμπειριών, να μπορούν να θέτουν από κοινού τις εμπειρίες που έχουν συσσωρεύσει. Είναι λοιπόν ένας τρόπος για να μπορέσουμε να προωθήσουμε περισσότερο το θέμα αυτό. Για τα εμβόλια, παραδείγματος χάρη, να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Συνάδελφε Ντορνάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Προέδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγό τη Διατλαντική Συμφωνία προβλέπουν να αποσυρθούν οι τελευταίοι φραγμοί τη ευρωπαϊκή οικονομία προστάτευαν από τι ωρέξει τη Αμερικανική αγορά. Δεν πιστεύετε ότι δεν είναι μόνο θέμα εμπορικό, αλλά είναι και θέμα υγεία και διατροφή. Λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια οι μεγάλοι όμιλοι αμερικανικοί προσπαθούν να κυριαρχήσουν στην ευρωπαϊκή γεωργία μέσα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των αδειών ευαισθητεχνία ή να πουλήσουν προϊόντα που αρνούμεθα μέχρι τώρα λόγω του ότι δεν συμμορφωνόταν με τι προδιαγραφέ μα όσον αφορά τη διατροφή και την ανεχνευσιμότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να δεχτεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντρίψει του γεωργού και του παραγωγού με απαιτήσει και προδιαγραφέ, αλλά θα δεχόταν ελαφρύνει τι όλε διατάξει ρυθμιστικέ για να ικανοποιήσει τι φιλοδοξίες ε, του τομέα των ελευθερών συναλλαγών. Πώς θα προστατεύσετε τα προϊόντα μας κύριε Επίτροπε και τη διατροφή μας απέναντι σε μια αμερικανική βιομηχανία που είναι λιγότερο συνετή όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Atsakydamas į klausimus anksčiau, aš jau išreiškiau labai aiškiai. Νομίζω ότι ήδη έχω δώσει μια απάντηση στο ερώτημά σας. Έχω τονίσει την θέση μου με σαφήνεια ως, ε, και ως επαγγελματίας του υγειονομικού τομέα αλλά και ως πολιτικός και ως αρμόδιος για την προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας. Τα πρότυπά μας δεν θα υποβαθμιστούν και ούτε θα πρέπει να παραγνωριστούν από την άλλη πλευρά. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, γίνουν υποδέστερα και οι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτά τα πρότυπα και να μπορέσουν να δώσουν αυτά τα πρότυπα και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζετε ότι τα πρότυπά μας είναι ιδιαίτερα υψηλά και εδώ είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να κυκλοφορούν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι μια προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε τόσο ψηλά λοιπόν πρότυπα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα δεχτούμε να υποσκαφθούν αυτά τα πρότυπα. Δεν είναι κάτι το οποίο επιδέχεται συζήτηση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια συμβαστική λύση που θα οδηγήσει σε, μείωση των προτύπων μας. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μικολάτσικ. είχατε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, Δόκτωρ Ανδριουκάητης, τα βλαστοκύτταρα, τα εμβριονικά, τα εμβρι... δεν έχουν ε, οδηγηθεί σε θεραπευτικές ε, αγωγές μέχρι τώρα, παρότι αυτό που πιστεύουμε. Είναι επίμαχο θέμα δεδολογικά, όμω παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τα εμβριακά αυτά βλαστοκύτταρα. Περίπου 2 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε ε, ζήτησαν να απαγορευτεί αυτή η έρευνα ε, κατόπιν δική μα πρωτοβουλία, ενό από εμά. Αγνοήθηκε όλη αυτή η κίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ποια είναι η δική σας επαγγελματική και προσωπική θέση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Εσείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσετε μια ανεξάρτητη έκθεση όσον αφορά τις ψευδείς υποσχέσεις για θεραπείες που βασίζονται στα ε, εμβριακά ανθρώπινα βλαστοκύτταρα. Και τέλος, προτίθεστε να ενισχύσετε προγράμματα με βλαστοκύτταρα ενηλίκων όσον αφορά ε, την μεγαλύτερη χρησιμοποίηση αυτών για θεραπευτικές αγωγές. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό το οποίο θέσατε και χαίρομαι που είστε συνάδελφος και του ιατρικού τομέα. Βλέπω λοιπόν ότι γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα αυτά. υπάρχει μια μελέτη για το θέμα του, της αποκωδικοποίησης του DNA και της δυνατότητας να χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιστημονικές γνώσεις για την θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Εδώ υπάρχει ένα ηθικό δίλημα το οποίο είναι σαφές και από αυτή τη μελέτη. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τα ζητήματα αυτά. Δεύτερον, είναι ορθό αυτό που είπατε, ότι η χρήση βλαστοκυτάρων για θεραπευτικούς στόχους, τουλάχιστον στις χώρες που γνωρίζω εγώ, έχει μέχρι στιγμής τύχη διαφορετικών ερμηνεών. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει προκύψει, παρά το γεγονός ότι έχουν δοκιμαστεί διάφορα και υπάρχει μια βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδος η οποία να έχει εξασφαλίσει την εγκυρότητα και να έχει θεωρηθεί ότι είναι μια θετική μέθοδος η οποία μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Εάν λοιπόν υπάρξει μια τέτοια μέθοδος η οποία να μπορέσει να εφαρμοστεί, αυτό θα είναι θετικό. Αλλά προς το παρόν πρέπει να δώσουμε εμείς μεγαλύτερη έμφαση στην ε, αντιμετώπιση, στην, μάλλον στην αξιολόγηση αυτών των μεθόδων. Και δεχούμε ότι έχετε δίκιο. Δυστυχώς βέβαια η έρευνα δεν είναι στον δικό μου τομέα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι καλύτερο να το θέσετε στον αρμόδιο επίτροπο για την έρευνα, αλλά αυτό που λέτε πιστεύω ότι είναι σωστό. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Πόξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άνδριου Κάιτης, εδώ είμαι πίσω σας. Είναι δύσκολο να με δείτε. Αναφερθήκατε στην επιδημία του ιού έμπολα στην αρχική σας ομιλία αλλά αντιμετωπίσουμε και μια επιδημία καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταλάβουμε το επίπεδο αυτής της ε, ε, ασθένειας έχουμε 150.000 άτομα που πεθαίνουν από καρκίνο του παχαίου σεντέρου και του ορθού κάθε χρόνο. Υπάρχει μεγαλύτερη λοιπόν θνησιμότητα για τον παγκρεατικό καρκίνο και για άλλες μορφές. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σαφή μηνύματα είναι σαφές ότι η απάντηση που έχουμε δώσει σε αυτά τα προβλήματα δεν ήταν επαρκή. Σε ποιο βαθμό ο καρκίνος και η αντιμετώπιση του θα είναι μία από τις προτεραιότητές σας και εάν ναι, τι ακριβώς θέλετε να προτείνετε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Αγγίξατε ένα πολύ οδυνηρό θέμα. Όχι μόνο ο καρκίνος, αλλά και τα καρδιακά νοσήματα, ενδοκρινικές ασθένειες. Όλες αυτές οι ασθένειες δημιουργούν μεγάλα προβλήματα και οδηγούν και στην γύρανση του πληθυσμού της Ευρώπης. 85% των, των ασθενειών των χρονίων ε, προέρχονται από αυτά τα προβλήματα και είναι μεγάλο βάρος για τους πληθυσμούς μας και για τις χώρες μας. Εάν ε, προσπαθούσαμε να τα φανταστούμε όλα αυτά από οικονομική σκοπιά, θα βλέπαμε ότι οι χρόνιες, οι οξύες, ε, χρόνιες ασθένειες είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν επιστημονικά μέσα πρόληψης βέβαια των ασθενειών αυτών. Όλοι γνωρίζουν ότι έγκαιρος εντοπισμός η, και η προφύλαξη, οι έγκαιροι, κυρίως στην περίπτωση του καρκίνου, αποτελούν λύση που πρέπει να ακολουθείτε. ποιο ποσοστό του πληθυσμού λαμβάνει προληπτικά μέτρα κατά του καρκίνου, του παχιός εντέρου ή του ορθού είναι πολύ μικρό. Μίλησα με ειδικού του τομέα της ογκολογίας και μου είπαν ότι θα μπορούσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο μέσω εφαρμογών ακόμα και στα κινητά τηλέφωνα. Θα μπορούσαμε να εφαρμόζουμε και προληπτικά προγράμματα, να ξέρει ο κόσμος ότι έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει να κάνει εξετάσεις σε κέντρα υγείας ότι είναι δυνατόν η πρόληψη να συμπεριλαμβάνει περισσότερους και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος χωρίς πρόληψη. Πρέπει να ασχολούμαστε με την πρόληψη και τη θεραπεία και με τις συνέπειες της ασθένειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ούτω ώστε να μπορέσει ο κόσμος να χρησιμοποιήσει την πρόληψη να πληροφορηθεί κατάλληλα μέσω τηλεόρασης, μέσω εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου. Πολύ συχνά βλέπω το κανάλι Euronews, δίνει πολλές πληροφορίες για τον καιρό στην Ευρώπη, αλλά ποτέ δεν λέει ποιο είναι το επίπεδο, τι προξενεί ο ήλιος και η δραστηριότητα του ηλίου. Και αυτό είναι σημαντικό για όσους έχουν προβλήματα δερματικά. Ευχαριστώ, The Messmaker. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφοι επίτροπε για το κόμμα μου είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη να φροντίσει να υπάρχει ποιοτική και επιστημονική φροντίδα υγείας. Οπότε δύο ερωτήσεις. Ε, μιλάμε για μια κατευθυντήρια γραμμή η οποία θα είναι evidence-based practice, ενώ κάποια κράτη-μέλη χρησιμοποιούν και εναλλακτική ιατρική. Τι άποψη έχετε για αυτή την διπλή προσέγγιση και για την ε, πιθανή αναγνώριση ή μη αναγνώριση αυτού, του, αυτής της ε, δυνατότητας. Επίσης, για το ότι η αρχή εποπτείας των φαρμάκων πήγε από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας με ανισχύ και εμένα όπως και τους συναδέλφους και η ερώτησή μου είναι τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της απόφασης. Για να απαντήσω την, στη δεύτερη ερώτηση θα προσπαθήσω εγώ η υγεία να είναι το πρώτιστο σε όλους τους τομείς. Ε, ο Επιτροπός Ανδρουκάητης, η κυρία Μπανκόφσκα, ε, Νίμιτσα, όλοι οι Επιτροποί, ε, η Επίτροπος η Αρμόδια για την Ανάπτυξη, όλοι, όλοι μας θα πρέπει να έχουμε κατά νου τις πτυχές της υγείας και να μας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Όταν μιλάμε τώρα για την υπηρεσία αυτή θα ληφθεί μία απόφαση από το Σώμα των Επιτρόπων την οποία εγώ θα πρέπει να εφαρμόσω όσον αφορά τώρα την εναλλακτική ιατρική και την αναγνώρισή της. Είναι βεβαίως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη κάνουν κάποια βήματα πρόοδου. Και η χώρα μου επίσης ε, συνέστησε μια ομάδα εργασία ε, και προσπαθεί να καταλήξει σε ένα νομοσχέδιο για την αναγνώριση της εναλλακτική ιατρικής, ε, τα ζητήματα υγείας, αξιοπιστίας, χρηματοδότησης. Κάποια βήματα γίνονται Λοιπόν, μπορούμε να ανταλλάξουμε βέλτιστες ε, πρακτικές και να προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε αυτά τα ζητήματα και νομίζω πως θα έχουμε συζητήσει και με τις εθνικές κυβερνήσεις ε, όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Μέισνερ, έχετε το λόγο. Κύριε Άντριου Κάιτης εδώ. Εγώ θα αναφερθώ σε κάποια ζητήματα που αφορούν το κάθε φίλο Θα προσπαθήσετε να σταματήσετε το να δηλώνονται ή διαφυλετικοί ως πνευματικά ασθενείς ε, σε διεθνή και εθνικά συστήματα και πώς θα φροντίσετε να υπάρξει παροχή υγείας συγκεκριμένα για τα άτομα αυτά. Dėkoju. σας ευχαριστώ. Και πάλι αυτό είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να τονίσω εδώ πέρα πως το πρώτο άρθρο της χάρτας ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ ωραία διατυπωμένο. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε κανένας είδους διάκριση, ειδικά στον τομέα της παροχής υγείας. Εδώ μιλάμε για τις υπηρεσίες υγείας, εδώ πρέπει να δούμε πως προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη υγεία. Ο όρκος Ιπποκράτη τα λέει αυτά. Και οι όρκοι άλλων επαγγελμάτων. Όλοι καταλήγουν στο ίδιο. Και η απάντησή μου είναι απλούστατη. Βεβαίω, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τα εθνικά συστήματα υγείας και πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως όμως όσα ισχύουν και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος Ροντρίγκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πορτογαλικά θα μιλήσω. Λόγω της ε, Τρόικα, οι λαοί της Ευρώπης οι λαοί μας δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που είναι ένα παγκόσμιο δικαίωμα. Είναι μια πραγματικότητα η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Τι θα κάνετε εσείς για να αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Έχετε το στόχο να κάνετε κάτι για να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Λοιπόν, για να πω την αλήθεια, αν σας κατανόησα σωστά, δεν κατάλαβα το πλήρες ε, θέμα, αναφερθήκατε στο ωκεάνιο, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι της ερωτήσεώς σας περί ιδιωτικοποίησεως των συστημάτων υγείας, αναφερόμενοι στους, στις περικοπές και στα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό είναι κάτι που έγινε με μηχανικό τρόπο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες πτυχές. Δεν μπορούμε να περικόπτουμε τον προϋπολογισμό υπονομεύοντας ε, τα δικαιώματα υγείας είτε είναι πρωτοβάθμια περίθαλψη είτε δευτεροβάθμια. Αν περικόπτουμε τον προπολογισμό, αυτό έχει οδυνηρές, πολύ οδυνηρές συνέπειες. Όταν μιλάμε λοιπόν για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας και την αντοχή τους, όταν αναφερόμαστε σε αυτό, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε κατά το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι να δώσουμε συμβουλές σε κάποιες χώρες όσον αφορά τα συστήματα υγείας και την περίθαλψη πρέπει να ελέγξουμε τι κάνουν οι χώρες, τι μέθοδο χρησιμοποιούν, ποια είναι η μεθοδολογία της ε, αξιολόγησης των συστημάτων υγείας, ούτω ώστε να μπορούμε πραγματικά να αποτιμήσουμε με συγκρίσιμο τρόπο τα 28 συστήματα υγείας αλλά οι καθολικές υπηρεσίες και η καθολική κάλυψη είναι ε, στο κέντρο των προσπαθειών. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις τεχνολογίες, την ηλεκτρονική υγεία, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, όσα εστιάζονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ε, ε, νοσοκόμους, ε, οικογενειακούς γιατρούς και πρέπει να καταλήξουμε όλοι μαζί σε κάποια πακέτα μέτρων και όλες οι προτάσεις θα πρέπει να τεθούν επί τάπητος. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρε Ζαβόρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Αντρουκάητης, εδώ είμαι, εδώ πίσω. Προτιμώ την ε, επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο κανονικά, αλλά θα επανέλθω στο θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και σύμφωνα με τη νέα προτινόμενη νομοθεσία η διασυνοριακή επιμόλυνση θα γίνει κάτι σημαντικότερο στο μέλλον με την ε, πρόταση αυτή. Εσείς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ζητήσετε υποχρεωτική διασυνοριακή συνορικά μέτρα κατά της επιμόλυνσης. Θα υποστηρίξετε το στόχο του Κοινοβουλίου για αυστηρά μέτρα ελέγχου και ούτω ώστε ο, ο, ε, ο ρηπαίνων εκείνος που μολύνει να πληρώνει και τα κάτι μέλη που δεν δέχονται τα γενετικά τροπημένους οργανισμού να μπορούν να κρατήσουν το, καθεστώ του, το καθεστώς τους που δεν δέχονται γενετικά τροποποιημένους οργανισμού, ακόμα αν και οι γειτονικέ τους χώρες έχουν εισαγάγει και έχουν εγκρίνει γενετικά τροποποιημένους οργανισμού. Ε, Σας ευχαριστώ λέει ο κύριος Κάρτης. Είναι προφανές αν μια χώρα επιτρέπει στους γεωργούς τους να καλλιεργούν <clears throat> προϊόντα γενετικά τροποποιημένα και μια άλλη χώρα δεν το δέχεται και τα, οι καλλιέργειες αυτές φτάνουν 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, φυσικά ο άνεμος μπορεί να φέρει την, ε, ε, τους σπόρους, την κόνη των ε, ανθέων κτλ στην άλλη χώρα και με τον τρόπο αυτό να υπάρξει μόλυνση από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο και πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους τους εμπλεκόμενους. Μπορούμε, πρέπει να εστιάσουμε στο θέμα του πώς μπορούμε να προστατεύσουμε ένα κράτος μέλος από ρήπανση που προέρχεται από τα σύνορά της από άλλες χώρες. Πρέπει να είναι ε, σίγουροι και οι καταναλωτές ότι έχει εξασφαλιστεί η υγεία τους στην περίπτωση αυτή. Αυτό είναι λοιπόν ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μόνο ένα τυφλό θα θεωρούσε ότι αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να σα δώσω μια συγκεκριμένη υπόσχεση για το αν τα μέτρα αυτά θα είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, αλλά σίγουρα θα συζητήσω το θέμα αυτό με όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί πρέπει να εξετάσουμε όλους τους μηχανισμούς οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Φυσικά όμως οι θέσει των κρατών μελών θα πρέπει να τύχουν σεβασμού και χώρε οι οποίε είναι όμορε μεταξύ του θα πρέπει να βρουν κάποια λύση για να εμποδίσουν μια τέτοια μόλυνση. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ. Η συνάδελφος Βενάντε Ζόμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Άντριου Γκάιτη, η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Εδώ είμαι ακολουθεί μια πατερναλιστική προσέγγιση μέχρι στιγμής. Θέλει να προστατεύσει τον καταναλωτή από τον εαυτό του. Και όχι μόνο με το αλκοόλ και τον καπνό, αλλά και στα τρόφιμα. Το βλέπουμε με τα διατροφικά προφίλ ε, του κανονισμού περί ισχυρισμών, οι οποίες τελικά καταλήγουν σε απαγόρευση διαφήμισης ε, τροφίμων που δεν αρέσουν στην Κομισιόν. Το πρόβλημα είναι πως ε, ε, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε μεμονωμένα τα τρόφιμα, πρέπει να δούμε την ετήσια πρόσληψη. Και το ερώτημά μου είναι, είστε διατεθειμένος να αποσύρετε αυτά τα διατροφικά προφίλ δεν ε, λειτουργούν, τεχνικά δεν στέκουν και πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ποιοι είναι οι ε, ορισμοί οι δικοί σας ε, όσον αφορά ακριβώς τον καταναλωτή και τον μέσο καταναλωτή, αν θέλετε, και τον υγιή καταναλωτή. Για να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από τις υποσχέσεις. Να υποσχόμαστε ξανά και ξανά. Εγώ νομίζω πως είναι καλύτερο να κάνουμε λιγότερα και να τα κάνουμε καλύτερα. Ειδικά στη δικιά μας τη δουλειά που υπάρχουν τόσα πολλά ζητήματα και προβλήματα πρέπει να παραδεχτώ πως ε, τα ζητήματα αυτά της σήμανσης είναι πάρα πολύ περίπλοκα. Είτε μιλάμε για ζάχαρη, οξέα, θερμίδες, ε, είναι δύσκολο το να βάλουμε κάποια ετικέτα, όπως διαφέρουν άλλωστε, όπως διαφέρει και η δίαιτα και η διατροφή του καθενός. Αν ένας ε, ασθενής πάει σε ένα γιατρό, ο γιατρός του δίνει μια ιατρική συμβουλή, μετά είναι επιλογή βεβαίως του ασθενούς, το καταναλωτή, ποια προϊόντα θα αγοράσει. Είναι περίπλοκο λοιπόν το ζήτημα. Εγώ δεν ε, θεωρώ πως ε, μπορώ να δώσω την τέλεια λύση. Πρέπει να το συζητήσουμε, οι απόψεις ε, διήστανται και δεν είναι τυχαίο το ότι η Κομισιόν καθυστερεί εδώ πέρα. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες λύσεις. Πρέπει να επιληθεί όντως το ζήτημα, αλλά το να σας δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή θα ήταν ανεύθυνο νομίζω. Σας ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Παρνιού έχει το λόγο. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω επί της καλλιεργίας γενετικά του οργανισμού και προχωρήσω πιο μακριά. Στις αρχικές σας ομιλίες και σε απάντηση του συναδέλφου Φρίντερ Κλίζε είπατε ότι όταν εκλεγείτε τον Νοέμβριο ε, θα ε, προωθήσετε το πακέτο και αναφερθήκατε στην αρχή της επικουρικότητας ότι θα γίνει σεβαστή και δεν θα συγκρουστείτε με τα κράτη-μέλη κάποιοι εμεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου λέμε ότι θα έπρεπε η κοινή θέση του Συμβουλίου να βελτιωθεί και να ενισχυθεί. Μπορούμε να έχουμε την υποστήριξή σας σε αυτή την προσπάθεια που θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινή θέληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 19 κράτη-μέλη ήταν αντίθετα όσον αφορά την καλλιέργεια γενετικά τροπεμένων οργανισμών, αλλά τελευταία χρόνια ασκήθηκαν κάποιε πιέσει για να επισημοποιηθεί κάποιε κάποιες αιτιολόγηση απαγόρευση που έχει πολλά και να συμφωνείτε μαζί μα Να καταρτιστεί κατάλογο ε, πιο σαφή όσον αφορά τι απαγορεύσει, να επιτρέπονται πιο περιοριστικά μέτρα για να αποφευθεί η μόλυνση από γειτονικέ περιοχέ που καλλιεργούνται γενετικά τροπεμένοι οργανισμοί και σύστημα αποζημίωσης των γεωργών που θα είναι θύματα της μόλυνσης και ε, αν θα γίνεται ε, κάποια αξιολόγηση του κινδύνου που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τροφίμων. Λοιπόν, αυτό θα ήθελα να επιβεβαιώσετε, ότι θα μας στηρίξετε. Πρέπει να αποδεχτώ ότι προσωπικά συμφωνώ με τη θέση που εκφράζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπόκειται στην επικουρικότητα. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο δοκιμάζει την ανεξαρτησία και την επικουρικότητα των κρατών μελών. Οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί προφανώς παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι δέσμοι μέτρων για τις ε, γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες κινείται με τον τρόπο αυτό. Πρέπει τα κρατημένα να καταλήξουν στις δικές τους αποφάσεις, θα είναι υποχρεωμένα να αναμείνουν τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα προερχέται από την Κομισιόν. Ακόμα και αν δεν συμφωνούν. Είναι λοιπόν μια παράξενη αντιπαράθεση και θα πρέπει να βρούμε και μια λύση για το θέμα αυτό. Για, στην δεύτερη ανάγνωση είδα να υπάρχει αυτή η τάση προς την κατεύθυνση των κρατών μελών. Τώρα, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με διαμεθοριακή μόλυνση των, επιμόλυνση των καλλιεργειών. Εδώ θα χρειαζόμουν περισσότερες επιστημονικές εμπειρογνωμοσύνες και αναλύσεις για το θέμα αυτό. Και ενδεχομένω η ιδέα που αναφέρεται είναι ορθή. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχω αρκετές πληροφορίες για το θέμα αυτό. Ενδεχομένω θα μπορούσα να επιστρέψω αργότερα για το θέμα αυτό. Αλλά είναι σαφές ότι το πρόβλημα αυτό υπάρχει, ότι είναι ένα αναπόφευκτο πρόβλημα για την ανεξαρτησία της ε, υπηρεσίας τροφιμικής ασφάλειας και τις τεχνικές ε, με ανάλυσής της. Έχω ήδη πει και στο παρελθόν για όλα αυτά τα θέματα είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Grazie. Σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος James Nicholson. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, υποψήφιε Επίτροπε. Συνεχίζεται το έβδομος γύρο γύρος των ε, συζητήσεων για την συμφωνία TTIP μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους πιο επίμαχους τομείς είναι αυτός που έχει να κάνει με την ε, εναρμόνιση στον φυτο-υγειονομικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι οι αγρότες Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παραμείνουν πιστοί στο υψηλότερο επίπεδο ε, προτύπων προστασίας για την παραγωγή ε, τροφίμων. Αυτά τα πρότυπα όμως δεν ακολουθούνται από άλλες χώρες και επιφέρουν ένα πρόσθετο κόστος για τους ε, γεωργούς. Εάν εγκριθείτε ως επίτροπος πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα διατηρηθούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα προστατευτούν οι τοπικοί καλλιεργητές και παραγωγοί και τώρα και στο μέλλον. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας και πράγματι νομίζω ότι ήδη έχω δώσει την απάντηση που επιζητείτε. Αυτό το οποίο, για το οποίο μπορώ να δεσμευτώ ενώπιον σας σήμερα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτώ να χαμηλώσει το επίπεδο των προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν αφορά μοναχά τα τρόφιμα, αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό, αφορά τα φαρμακευτικά σκευάσματα κτλ. Δεν βλέπω καμία δυνατότητα να υπάρχει συμβαστική λύση ή άλλη διέξοδος για μας. Όλα αυτά φυσικά εμπλέκονται σε ένα σύνολο θεμάτων γιατί έχουν να κάνουν και με την υγεία των καταναλωτών, με το μέλλον των παιδιών μας Είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις μελλοντικέ αυτές γενιές, οι οποίες θα αναλάβουν τη σκητάλη από μας και είμαστε επίσης και υπεύθυνοι για την ε, τον αγροτοτροφημικό κλάδο στην Ευρώπη και την απασχόληση στον τομέα αυτό. Είναι ένας τομέας ο οποίος δημιουργεί τεράστια προσθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν πρόκειται λοιπόν για τα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, αυτά είναι ακρογωνία λήθος για την επιτυχία του αγροτοτροφημικού τομέα και είναι εδώ πιστεύω απόλυτα σαφής η θέση της Κομισιόν, όχι σε οποιαδήποτε υποβάθμιση των προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι Χουιτέμα για το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ υποψήφια επίτροπε. Το όλο συνέστημα στην Ευρώπη για τα γενετικά τοπιμένα τρόφιμα είναι πολύ αρνητικό. Ε, η καινοτομία στο γεωργικό τομέα βλάπτεται. Θα μπορούσαμε όμως να βελτιώσουμε την κατάσταση μειώνοντας τα φυτοφάρμακα. Ε, υπάρχει και στην Ολλανδία μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, καταπολέμονται τα φυτόφτερα που είναι μια ασθένεια των, των γεωμήλων και μπορεί να μειωθεί κατά 50% σε κατά κάτι μέλη με τη χρήση των σωστών γεννήτικων. Δεν χρησιμοποιούμε γονίδια από άλλα είδη, αλλά μεταφορά γονιδίων στο ίδιο είδο. Η ΕΦΣΑ ήδη το 2012 συνεπέρανε ότι αυτό το σύστημα είναι πολύ σωστός τρόπος και αναπαραγωγής των φυτών και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι γενετικά τροπημένος οργανισμός. Οι νέες τεχνικές αναπαραγωγής των φυτών πιστεύετε ότι τελικά κρίνονται βάσει συναισθημάτων και όχι επιστημονικών στοιχείων και ότι αυτό είναι κάτι που εμποδίζει την αντιδότηση των τεχνικών. Υποψήφιος Επίτροπο συμφωνεί ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ανοιχτή σε νέε μεθόδου αναπαραγωγή φυτών που μπορεί να είναι κάτι επωφελέ και για του καταναλωτέ και για το περιβάλλον και πότε αποφασίζει να αποκλείσει το Sys Genesis από τον κατάλογο των απαγορευμένων αυτών τεχνικών που θεωρούνται ότι αποτελούν γενετική τροποποίηση τόσο ώστε αυτή η επωφελής μέθοδος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. E, να σας πω την αλήθεια. Έτσι για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακριβώς ε, και τις αρμοδιότητες για να εφεύρω εγώ γενετικά τροποιημένες ποικιλίε. Αλλά και η επιλογή που γινόταν ε, επί 300 χρόνια ακριβώς οδηγεί στο να καλλιεργούνται οι πιο ανθεκτικές ποικιλίε. Ε, το ίδιο και με τα ζώα τα τελευταία 500 χρόνια μέσω της επιλογής ε, ε, κάποιες ποικιλίε. Πώς θα το κάνουμε αυτό τεχνητά. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ναι. ε, επιστημονικά στοιχεία. Αλλά ε, τώρα πειράματα με τη φύση ε, δημιουργούν ζητήματα ηθικής ε, και ζητήματα ασφαλείας. Εγώ είμαι ανοιχτός στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, αλλά πάντα βασιζόμενοι σε στέρεες επιστημονικές βάσεις. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος Φορέντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσουμε για την προστασία της υγείας σημαίνει επίσης και προστασία της υγείας και της ασφαλείας των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα των εργαζομένων των μεγάλων βιομηχανιών για να αποφύγουμε να υποστούν βλάβη στην υγεία και επίσης να μην βλάπτονται την οι κοινωνικοί πληθυσμοί. Μιλώ για μια υπόθεση της Σύμβασης στο Τάροντο. εκεί υπάρχει μεγάλη βιομηχανία για την παραγωγή χάλιβα όπου εκεί είχαμε εντυπωσιακά στοιχεία όσον αφορά τον θάνατο εργαζομένων και βλάβες για το περιβάλλον. Αυτή η κατάσταση οδήγησε το 2012 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει η διαδικασία παράβασης κατά του Ιταλικού κράτους που δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ε, ζητώ, ποια πρωτοβουλία προτίθεστε να αναλάβετε για να ε, προστατεύσετε το περιβάλλον και την υγεία. Προτίθεστε να προβλέψετε νέες διαδικασίες για κυρώσει ad hoc, για να επιβάλλετε οι ίδιοι εκείνοι που χειρίζονται τις εγκαταστάσεις του δημόσιου ιδιωτικού τομέα να ε, λάβουν τα μέτρα, τα αναγκαία για να αποφευθεί μόνιμη βλάβη της υγείας των πολιτών. Και οι πολίτες αντί να πρέπει να πληρώνουν τελικά οι ίδιοι πολίτες μέσω του κράτους τις βλάβες που υπο, ε, στις οποίες υπόκεινται οι ίδιοι αλλά και τις βλάβες του περιβάλλοντος. Κοιτάξτε, το σύστημα αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την Ιταλία αλλά για πολλά κράτη-μέλη και γεγονός είναι πως οι ε, ειδικοί της ασφάλειας και της υγιεινής ε, στην εργασία ε, που αναλύουν το χώρο εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντική και υπάρχει έλλειψή τους στα κράτη-μέλη. Νομίζω υπάρχουν και συλλογικές ε, συμφωνίες οι οποίες θα έπρεπε επίσης οι συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων να προβλέπουν και κάτι για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστιες ε, διαφορές ε, η κοινωνική χάρτα επίσης θα πρέπει να αναφέρει κάτι και με αυτό το έγγραφο πρέπει να κινηθούν τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουμε μία βάση σε αυτό το τομέα. βεβαίω υπάρχουν οι αρμοδιότητες των κρατών μελών αλλά και οδηγίε, οι οποίες παραβιάζονται και διαδικασίες σε παραβάση. Από τη σκοπιά λοιπόν της πολιτικής υγείας εγώ θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Αλλιώς δεν θα σέβομαι και το επάγγελμά μου. Είναι σαφές λοιπόν πόσο μπορούμε να δούμε αυτά τα ζητήματα σε μεγάλη λεπτομέρεια. δεν ξέρω συγκεκριμένα τι σημαίνει στην Ιταλία, αλλά είναι σημαντικό το ζήτημα, θα με απασχολήσει. Σας ευχαριστώ, συνάδελφος Σλοβέν. Ευχαριστώ, θα μιλήσω σου ειδικά. Εδώ κάθομαι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει <clears throat> εντοπίσει ε, την αντίσταση στα αντιβιωτικά, την των μικροοργανισμών ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τη δημοσία υγεία και εδώ θα πρέπει να δράσουμε με ταχύτητα εάν δεν θέλουμε να υπάρξει ένα μεγάλος, ένας μεγάλος αριθμός θανάτων στην Ευρώπη από ασθένειες. Υπήρξε ένα σχέδιο δράσης το οποίο ξεκίνησε το 2011 από την Κομισιόν για να αντιμετωπίσει το θέμα της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην ρίζα του, γιατί όλο και περισσότερο παρέχονται περισσότερα αντιβιωτικά στα ζώα τα οποία είναι ασθενή και στα άτομα, στους ανθρώπους. Υπάρχει λοιπόν ε, αδιάκριτη χρήση των ε, αντιβιωτικών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ιταλία και στην Κύπρο, παραγωγός χάρη, υπάρχει τεράστια χρήση αντιβιωτικών επίσης και στα ε, στην εκτροφή χείρων στη Δανία έχουν εμφανιστεί οι βακτηρίδια τα οποία αντέχουν σε όλες αυτές τις μορφές αντιβιωτικών και αυτό διοίκησε σε ανθρώπινους θανάτους. Πώς λοιπόν θέλετε να εφαρμόσετε αυτή την οδηγία για τη χρήση των αντιβιωτικών στην κτηνοτροφία. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν μια νέα ε, οδηγία για την ευζοία των ζώων, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, Ανδρίου Κάιτης. Έχει δύο πτυχές αυτό το ερώτημα. Από τη μία πλευρά η αντίσταση στα αντιβιωτικά των μικροβίων και των μικροοργανισμών και δεύτερον το θέμα της προστασίας των, της υγείας των ζώων. Ξεκινώ με το πρώτο θέμα. Το ότι πράγματι γίνονται πάρα πολλά, πολύ μεγάλη χορήγηση αντιβιωτικών από τους κτηνιάτρους είναι γεγονός και δεν πρέπει να δίδονται για προφυλακτικούς λόγους τα αντιβιωτικά, αλλά μόνο για την καταπολέμηση ασθενειών. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρης ε, επαγρύπνηση και εποπτεία. Δεν μπορούν να δίδονται αντιβιωτικά παρά μόνο όταν είναι άρρωστο το ζώο. Το θέμα τώρα της αντίστασης στα αντιβιωτικά και για τους ανθρώπους υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Έχω δει και εγώ στην πράξη ως ιατρός ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο έλεγχος για τα αντιβιωτικά όταν χορηγούνται σε ανθρώπους <clears throat> και όχι μόνο στα νοσοκομεία αλλά και σε καθημερινό επίπεδο. Είναι δραματικό πόσοι οι άνθρωποι στην Ευρώπη πεθαίνουν πια χιλιάδες που έχουν χάσει την αντίστασή τους στις ασθένειες και μπορούν σε ένα νοσοκομείο να, πάρουν μια, να κολλήσουν μια ασθένεια γιατί οι μικροοργανισμοί είναι ανθεκτικοί πια στα αντιβιωτικά. Πρέπει λοιπόν το σύστημα το υγειονομικό μας να τροποποιηθεί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών σε αντιβιωτικά. Φυσικά το θέμα αυτό όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και το οποίο αφορά και, τους, και την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων. Είναι ένα τεράστιο λοιπόν πρόβλημα και εγώ ως ιατρός, ως επαγγελματίας γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα αυτά. Για την ε, ευζοία τώρα των ζώων και την ομοθεσία στον τομέα αυτό δεν θέλω να σας δώσω εδώ μια υπόσχεση αλλά εγώ είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό και να το λύσω. Σας ευχαριστώ συνάδελφος Μπάλτσο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αντρουκάιτε. Η πολιτική όσον αφορά την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει όλη, όλη την αλυσίδα διατροφής. Συμπεριλαμβάνονται και γενετικά τροπημένοι οργανισμοί. Η οδηγία στην Ευρώπη σε τι πρέπει να βασίζεται. Στην εσωτερική αγορά πρωτίστως ή στην προστασία του περιβάλλοντος. Ποιος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος, ποιος αποτελεί προτεραιότητα. Μόνο ένας παράγοντας μπορεί να είναι σημαντικότερος από τον άλλον. Ερώτηση 2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είπε το εξή ότι η χρήση τεχνικών που δεν βασίζονται σε γενετικά τοπιμένους οργανισμούς ή βιώσιμες επενδύσεις σε βιώσιμη εντατική γεωργία, βάσει αυτών μπορεί η Ευρώπη να γίνει κυρίαρχη στην αγορά αυτό ε, δεν ισχύει για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εσείς με ποια πλευρά είσαστε. Με την άλλη πλευρά που ακούσατε α, προλίγο από τον συνάδελφο ή στην άλλη πλευρά. Το kontekstą, bet ε, ε, Ακούστε με... Ίσως δεν κατάλαβα καλά το πλαίσιο της ε, ερώτησης, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω. Προσπαθώντας ε, πρώτα απ' όλα να πω το πού στέκομαι εγώ. Εάν δούμε σήμερα την κλιματική αλλαγή, αν δούμε τις ε, εντάσεις στο φυσικό περιβάλλον, τη μείωση της βιοπικιλότητας σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπουμε επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία. Εγώ συμμετείχα και στη Γενική Συνέλευση του ΠΟΗ, Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, και εκεί πέρα αναλύθηκε η σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και ανθρώπινης υγείας. Ζούμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον Τώρα το ποια πτυχή είναι πιο σημαντική, νομίζω η απάντηση εδώ πέρα είναι σαφής. Η προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς αυτό δεν υπάρχουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Το μιλάμε τώρα για τα γεωργικά προϊόντα, τους τρόπους παραγωγής, ε, τη βιολογική καλλιέργεια. Πρέπει να βρουν τη θέση τους ε, στην αγορά. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για εντατική καλλιέργεια αν και βεβαίως πρέπει και αυτή να τη δούμε. Πρέπει να υπάρχουν και βιολογικά προϊόντα π.χ. στα σχολεία. Αυτό είναι κάτι το ε, επενετέ οπωσδήποτε και είναι αρμοδιότητα όμως των καρτόμελων Τώρα δεν μπορώ να σας πω σαφώς αν ανήκω σε μία από τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ κυρία Ντελάη. Σα σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, εδώ είμαι. Μπροστά σας, κατευθείαν μπροστά σας. Υπάρχει η κατασπατάληση των τροφίμων που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και αυτό ε, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στην ιδέα της κυκλικής οικονομίας. Μήπως μπορείτε να μας διευκρινίσετε ποιε είναι οι δράσει που θα αναλάβετε για να αντιμετωπίσετε τη σπατάλη των τροφίμων και τι θα κάνετε και μέσα στα πλαίσια της αντιμετώπισης στον τομέα της γεωργίας. Είσαστε έτοιμο να υποστηρίξετε μια ευρωπαϊκή κοινή δράση για την συλλογή από τους ε, παραγωγούς και ε, της διανομή της ανθρωπιστικές και φιλανθρωπικές οργανώσεις ε, οποροκυπευτικών και άλλων προϊόντων που είναι απαραίτητες απαραίτητα για την ισορροπία της διατροφής. Επίσης το θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών. Είναι ένα θέμα το οποίο καλύπτεται ήδη από διάφορα νομοθετήματα, αλλά υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για βελτίωση. Εσείς ως αρμόδιος επίτροπος για την τροφιμική ασφάλεια προβλέπετε να αναλάβετε δράση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Αντριο για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες έχω ήδη εκφραστεί. Θα πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες προσπάθειες και να καταλήξουμε σε πιο σαφή κριτήρια για τον καθορισμό των ενδοκρινικών ε, διαταρακτών ώστε να αποκλείσουμε οποιαδήποτε βλάβη προς το περιβάλλον και προς την ανθρώπινη υγεία. Για την απόρριψη τώρα και τη σπατάλη Βλέπετε εδώ πέρα αυτό το μπουκαλάκι. Έχει μια ημερομηνία ε, λήξης το μπουκαλάκι αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το πίνω αυτό το νερό μέχρι ε, τον επόμενο μήνα ή όχι. Δεν υπάρχει σαφήνεια Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια μεγαλύτερη κατανόηση από τον καταναλωτή αν αυτό πρέπει να το πιει ή να το πετάξει. Τι σημαίνει αυτή η ημερομηνία λήξη σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές ότι μπορεί ακόμα να καταναλώσει αυτό το νερό και μετά την υποτιθέμενη αυτή ημερομηνία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για τους καταναλωτές και εδώ χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή με τους παραγωγούς ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη κατασπατάληψη, κατασπατάληση προϊόντων τα οποία απλώς πετιούνται γιατί έχει περάσει μια ημερομηνία καταληκτική. Αυτό είναι λοιπόν απαραίτητο. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος Βίλμοντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Τον περασμένο Δεκέμβρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξεπώνησε έκθεση για την εκκλησία για τη χώρα προέλευση όσον αφορά τα μεταποιημένα τρόφιμα και το κρέα. Είπε ότι οι καταναλωτέ θέλουν την επισήμανση, αλλά είναι πάρα πολύ δαπανηρή. Δυστυχώ αυτό βασιζόταν με ίδιε εκθέσει τη βιομηχανία και έρευνα καταναλωτών στη Γαλλία κατέδειξε ότι η εκθεσία όσον αφορά τη χώρα προέλευση κρέα σε έτοιμη μπολονέ κοστίζει λιγότερο από ένα σεντ. Δηλαδή πολύ χαμηλή τιμή. Οι καταναλωτέ απαιτούν τίμιε πληροφορίε, ειλικρινεί πληροφορίε για την προέλευση του κρέατο, διότι είχαμε και το σκάνδαλο του κρέατο αλόγου εδώ και ένα χρόνο. Θα προτείνεται νομοθεσία για την ετικετοθεσία και την ανείχνευση του κρέατο, την προέλευση. Και επίση περιμένουμε και για το αλκοόλ και Οι καταναλωτέ θα πρέπει να θέτουν τι πληροφορίε ούτω ώστε να κάνουν επιλογέ υγιεινέ. Όπω πόσε θερμίδε ε, ε, βρίσκονται εντό του αλκοολούχου ποτού, ε, πότε να περιμένουμε την πρόταση νομοθεσία και θα ενταχθεί και το ενόπνευμα στο ίδιο πλαίσιο όπως και τα άλλα τρόφιμα για να σταματήσει η σύγχυση. Λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο το 2007 διάφορα προφίλ διατροφικά και περιμένουμε ακόμα κάποιες πληροφορίες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Eh, Όσον αφορά λοιπόν αυτά τα προφίλ τα διατροφικά που αναφέρατε, είναι περιπλοκότατο ζήτημα που σχετίζεται με διάφορες διέτες, διάφορες ε, ε παραδόσεις και διάφορες παραδόσεις χωρών. Σε κάποιες χώρες τρώμε αλάτι και ψωμί, αλλού τρώνε περισσότερο τυρί. Κάποιες χώρες ε, ε, στηρίζουν ε, περισσότερο το καπνιστό κρέας, ε, το ζαμπόν το καπνιστό που έχει πολλά μπαχαρικά και εκεί ε, έχουμε ψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Είναι περιπλοκότατο το όλο ζήτημα και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το χρόνο της. Προσπαθεί να βρει λύσεις γιατί υπάρχουν δυσκολίες. Θα πρέπει να εξετάσω ενδελεχώς το ζήτημα. Τώρα η ετικετοθεσία και πληροφορίες όσον αφορά τις θερμίδες αλκοολούχα ποτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε εξαιρέσει για τους παραγωγούς ενοπνευματοδών ποτών. Η παραγωγή των ενοπνευματοδών ποτών ε, βάζουν το έτος παραγωγής στην ετικέτα και πράγματα που είναι θετικά για αυτούς. Αλλά οι θερμίδες δεν αναφέρονται καθόλου. Και είναι αρκετές οι θερμίδες στα αλκοολούχα ποτά, οπότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί. Επίσης, Α, το πρώτο ερώτημα μπορείτε να το επαναλάβετε, το πρώτο τμήμα της ερώτησης. Η χώρα προέλευσης για το κρέας στα μεταποιημένα τρόφιμα. Αυτή ήταν η ερώτηση. Απάντηση του υποψηφίου επιτρόπου. Γνωρίζω ότι πριν την ακρόαση μάλιστα, ήμουνα σε επαφή με τους διάφορους ειδικού και εξέτασα διάφορα στοιχεία. Και είδα ότι οι καταναλωτές μας ενδιαφέρονται, θέλουν να γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης, άρα πρέπει να το επανεξετάσουμε αυτό και να δούμε τι κόστος συνεπάγεται και ποιος πρόκειται να το πληρώσει και να καλύψουμε το κόστος. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε κάποια απάντηση. Ευχαριστώ, η συνάδελφος Γκίρλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να επανέλθω στους ενδοκρινικούς διαταράκτες και θέλω να τονίσω ότι αυτό πρέπει να είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές σας όπως είναι και της δικής μας Επιτροπής. Δεν ακούσαμε από εσά ακριβώς πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό πέραν του ότι είπατε ότι είσαστε έτοιμος να εξετάσετε και πάλι τα κριτήρια για το να χαρακτηριστεί μια ουσία διαταράκτης. Να σας ρωτήσω και πάλι σαφώς. Μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο κριτηρίων για να καθορίζετε τι αποτελεί ενδοκρινικό διαταράκτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση θα λάβει και υπόψη της την, ε, τον κίνδυνο έκθεσης σε τέτοιους διαταράκτες. Ναι, λέει ο κύριος ε, Κάιτης όταν γνωρίσω καλύτερα τον φάκελο αυτό, μάλλον όταν ήρθα σε επαφή με αυτό το φάκελο, κατάλαβα γιατί υπάρχει αυτή η προβληματική και γιατί ξεκινάει με τα προϊόντα καλλιντικών, με τα, τις συσκευασίε, με τα παρασιτοκτόνα και άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και, της, ε, και στην κτηνοτροφία. Είναι ένα πολιτικό πρόβλημα οι έρευνες που γίνονται τώρα καλύπτουν ένα ευρύ Ο τελικός κατάλογος κριτηρίων θα πρέπει να εγκριθεί λαμβάνοντα υπόψη όλες τις πτυχές και θα πρέπει να ακούσω και την άποψη των εμπειρογνωμόνων και των ειδικών για τον κατάλογο αυτό. Είμαι έτοιμος να επανέλθω λοιπόν στο θέμα αυτό από τη στιγμή που θα έχω όλες τις απαραίτητες γνώσεις. Θα ήταν ε, από τη δική μου πλευρά ανέθυνο να σας δώσω τώρα μια απάντηση χωρίς να έχω μπει σε βάθος στα θέματα αυτά. Είναι προφανές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα πολύπλοκα χαρακτηριστικά αυτών των ουσιών. Διαβάζω τι απαντήσει, κύριε Αντρουκάητη, του ερωτηματολογίου που λάβατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τα χαρά είδα ότι μία τη προτεραιότητέ σα θα είναι υποστήριξή σα καινοτόμων ε, συστημάτων υγείας, ούτως ώστε να είναι ισότιμη η περίθαλψη όλων των πολιτών και ταυτόχρονα τα συστήματα να είναι οικονομικά βιώσιμα. Θα τα στηρίξετε. Η δημόσια συζήτηση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας σχετίζεται άμεσα με θέματα δημοσιονομικά και τις τιμές των καινοτόμων φαρμάκων. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι καινοτόμες θεραπείες βελτιώνουν τα αποτελέσματα όσον αφορά την υγεία και συνεπιφέρουν και έμεσα ωφέλη όπως η οικονομία όσον αφορά τα συστήματα υγείας και τη κέρδη παραγωγικότητας. Εν γέννη, άνηση πρόσβαση σε καινοτόμε θεραπείε είναι πολύ σημαντικό θέμα και συζητείται σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και στη δική μου. Τι θα κάνετε ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα ωφέλη λόγω επενδύσεων στην υγεία θα λαμβάνονται σωστά υπόψη στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και τις συστάσεις που θα πορεύσουν και τι πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη προσέγγιση, πρόσβαση ε, των ασθενών στα αποτελέσματα τα θετικά όσον αφορά την υγεία τεχνολόγιας. Οι καινοτόμες ε, θεραπείες ε, και τεχνολογίες πρέπει να εξελογηθούν Με τις ε, κατάλληλες μεθόδους. Βεβαίως η καινοτομία κοστίζει και πρέπει μετά να ρωτήσουμε τη βιομηχανία γιατί, ε, γιατί βάζετε αυτή την τιμή στην καινοτομία. Αλλά πρέπει να υπάρχει καινοτομία και κάποιες επιτροπές να αξιολογούν την καινοτομία. Ε, υπάρχουν αυτές οι επιτροπές στα κράτη-μέλη, αλλά υπάρχει πρόβλημα με τη μεθοδολογία της αξιολόγησης. Πρέπει να υπάρχει ενιαία μεθοδολογία, είτε μιλάμε για τη Λιθουανία, τη Ρουμανία ή την Ισπανία. Πρέπει να συμφωνήσουμε για την αξιολόγηση της ε, καινοτομίας. Όταν μιλάμε τώρα για την οικονομική πτυχή βεβαίως, Έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης ε, των φαρμάκων ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Από πρακτική πείρα μπορώ να σας πω πως ε, μπορούμε να ε, κάνουμε οικονομίες ε, μέσω της καλύτερης ρύθμισης των γενώσιμων φαρμάκων. Να εξοικονομήσουμε δεκάδες της εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μετά μπορούν να πάνε σε ένα κοινό ταμείο και να συμφωνήσουμε που θα επενδύσουμε και να συμφωνήσουμε τη βιομηχανία ότι θα επενδύσουμε αυτά τα λεφτά στην καινοτομία και θα δεσμευτεί και η βιομηχανία σχετικά. Μπορούν να γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Βεβαίω υπάρχει και η επικουρικότητα των κρατών μελών και δεν μπορεί να τα επιβάλλει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πρέπει να λυθεί το ζήτημα. Ευχαριστώ, συνάδελφος Παουλούτσι έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ο κ. Πρόεδρος έχει δίκιο. Αυτές οι σπατάλες ε, των τροφίμων είναι ντροπή. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη σπαταλώνται 180 ε, κιλά τροφίμων ανά άτομο. Το 2020 αυτό θα αυξηθεί κατά 40%. Η παχυσαρκία τώρα πλέον είναι μεγάλη πληγή. Η παχυσαρκία ενώ ένα δισεκατομμύριο άτομα πεθαίνουν από την πείνα. Έχουμε τη μία πλευρά γη και νερό ε, σαν πόρους ε, περιορισμένους πόρους και από την άλλη πλευρά έχουμε μεγάλες πατάλες και δεν έχουμε πολιτική δράση. Λοιπόν, καλές οι πρωτοβουλίες, ε, οι φιλανθρωπικές, αλλά θα πρέπει η Ευρώπη να κάνει περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, σας θέτω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η δημοσίευση της ανακοινώσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μπλοκαριστεί όσον αφορά τη δημιουργία συστήματος ευρωπαϊκού βιώσιμου για επισητιστικού βλέπω να παίζει αποφασιστικό, βλέπετε να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην πολιτική σας πρωτοβουλία. Θα παρουσιάσετε σύντομα αυτή την ανακοίνωση σαν οδικό χάρτη για συγκεκριμένες δράσεις. Δεσμεύετε να προωθήσετε προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με ενοποιημένη προσέγγιση ε, τέτοια μεγάλα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ε, δεν υπάρχει αμφιβολία πως όταν μιλάμε για τα τρόφιμα που σπαταλάμε ε, τα γεγονότα είναι πράγματι επέσχυτα. Πρόκειται για ανεύθυνη διαχείριση πόρων και πρέπει να ληφθούν ε, μέτρα. Εγώ θα κοιτάξω την ανακοίνωση αυτή και την αναθεώρησή της και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι βεβαίως να αναθεωρήσουμε όλους τους κανονισμούς, τις ανακοινώσεις να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τώρα κάτι για τις νομοθετικές ε, προτάσεις ε, γιατί όπως είπα εργαζόμαστε συλλογικά στην Επιτροπή, αλλά οπωσδήποτε οι συζητήσεις θα είναι ανοιχτές μεταξύ της Κομισιόν και της ε, Επιτροπής σας και θα εξετάσουμε όλες τις σχετικές στοιχείες και σας διαβεβαιώ πως θα εργαστώ εντατικά. Σας... σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων που θα υποβληθούν από τους συναδέλφους της Επιτροπής Άγκρη. Ξεκινώ μέσω δίνοντας το λόγο στο συνάδελφο Herbert Dorfman. Η επίτροπε, εδώ είμαι. Έχω μια ερώτηση στον τομέα της υγιεινής. Ήδη από το 2007 είχε υποβάλει η Κομισιόν μια πρόταση για μικροεπιχειρήσεις με κάτω των 10 υπαλλήλων και το πώς θα τους ε, απελευθερώσει από την ε, γραφειοκρατία ειδικά όσον αφορά τον τομέα του ΧΑΣΠ παρόλα αυτά δεν πέρασε ποτέ αυτή η πρόταση από το Συμβούλιο παρά το ότι ε, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να υπάρξει μια απαλλαγή απλοποίηση του συστήματος χάσπη για τις επιχειρήσεις αυτές. Τι θα κάνετε εσείς για αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, η απαιτήσει ε, υγιεινής είτε μιλάμε για μικρές είτε για μεγάλες εταιρείες ε, πρέπει να ισχύουν. μια φορά μια μικρή εταιρεία τριών ατόμων φτιάχνει ξέρω εγώ φαγητό για έναν υπηαγωγείο. εάν ε, δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφές ε, θα δηλητηριαστούν τα παιδιά. Αν μια γυναίκα ας πούμε, που δουλεύει στην κουζίνα έχει ε, μια μόλυνση και επιμολύνει όλο το φαγητό με το σταφυλόκοκο. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για χαμηλότερες απαιτήσει. Άλλα πράγματα μπορούμε να τα δούμε. Υπάρχει νομοθεσία που συχνά αλληλεπικαλύπτεται. Ίσως σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε μια λογική λύση. Αλλά όταν μιλάμε για υγιεινή και προδιαγραφές, είναι ανεύθυνο να τις ε, χαμηλώσουμε. Η χώρα στην οποία κατάγομαι είχε περιπτώσεις με θανάτους παιδιών ακριβώς από την περίπτωση που ανέφερα. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η συνάδελφος Τζουφρίτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ήρθατε Επίτροπε, εδώ είμαι. Υπογραμμίσατε το ότι η υγεία είναι ένα αγαθό της κοινωνίας και θα πρέπει να βελτιωθεί αποτελεσματικότητα και η πρόληψη στον τομέα. Όπως γνωρίζουμε υπάρχει πολύ στενή σχέση μεταξύ της ευζοίας των ζώων και της ανθρώπινης υγείας. 70% των μολυσματικών ασθενειών είναι κοινέ μεταξύ ανθρώπων και ζώων δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν ότι η προστασία των ζώων στις εκμεταλλεύσεις είναι στεμιλιώδης αξίας. Πώς θα συμπεριφερθείτε όσον αφορά μελλοντικά μέτρα για την πρόθεση των καλών πρακτικών στον τομέα της κτηνοτροφίας. Ήδη αναφερθήκατε στο πόσο είναι αναγκαίο να γίνεται πιο υπεύθυνη χρήση των φαρμάκων και των αντιβιωτικών Πώς θα δράσετε όσον αφορά μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν τρίτες χώρες που επηρεάζουν και τη δημόσια υγεία και τον αθέμητο ανταγωνισμό και να αντιμετωπίσετε αιστείες ζωνώσεων που έχουν μεγάλο αντίκτυπο όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τέλος πάντα στο πρέγμα της ε, υγείας των ζώων ποια μέτρα θα αποφύγουν στο μέτρο του δυνατού το να υποφέρουν τα ζώα τη στιγμή της σφαγής τους. Taip iš tiesų. Πράγματι λέει ο κύριος Αντζήγου Κάιτης, τα ζώα, τα ζώα υποφέρουν πολύ συχνά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους ή κατά τη διάρκεια της φαγής τους. Στην περίπτωση της φαγής υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που βασίζονται στις θρησκευτικέ πεπιθήσεις που θα πρέπει να τις σεβαστούμε. Υπάρχουν συγκεκριμένες θρησκευτικέ παραδόσεις για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, η ευζοία των ζώων είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα για μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τρίτες χώρες, όταν ε, ετοιμαζόμουν για την ακρόαση αυτή, συζήτησα το ζήτημα αυτό με τους συναδέλφους μου γιατί με ενδιέφερε πάρα πολύ και ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι έμαθα ότι οι επιθεωρήσεις των κτηνιάτρων μας μπορούν να γίνονται και σε τρίτες χώρες που θέλουν να εξάγουν προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλιώς να εμποδίσουν τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων τους αυτών. Όταν μιλάμε για λοιμώδεις νόσους ή επιζωοτίες που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή τροφίμων, πρέπει να ξέρουμε ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρξει ε, εμποδισμό της ε, εισαγωγής των προϊόντων. Σε καμία περίπτωση οι χώρες δεν μπορούν να φέρουν επιζωτίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες. Ξέρουμε ότι είναι σαν τις πυρκαγιές οι, οι, οι ασθένειες και οι επιδημίες στον κόσμο μας και δεν έχω αρκετό χρόνο για τα αντιβιωτικά να σας επανέλθω, αλλά είμαι έτοιμο να συζητήσω μαζί σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τον έχει η συνάδελφος Πάουσαν. Εδώ είμαι κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας. Θέλω να επαναλάβω δύο δηλώσεις που έχουν κάνει οι προηγούμενοι ομιλητές. Πρώτα απ' όλα για το θέμα της χρήσης των αντιβιωτικών το γεγονός ότι τα δύο τρίτα όλης της χρήσης αντιβιωτικών γίνεται στην κτηνοτροφία και κυρίως για προφυλακτικούς λόγους γιατί δεν ξέρουν πια οι κτηνοτρόφοι πώς να, προσε... να προσέχουν τα ζώα τους πια και να τα εκτρέφουν σωστά. Οι περισσότερες από τις αστόνιες αυτές λοιπόν προέρχονται από τα ζώα που αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει και στο παρελθόν να δει από την Κομισιόν μια πρόταση για να υπάρξει γενική νομοθεσία που να αντιμετωπίσει την ευζοία των ζώων. Η Κομισιόν έχει δεχτεί μέσα στη στρατηγική της για την προστασία των ζώων αυτή την πρόταση. Και επομένως το ερώτημα προς εσάς είναι το εξής, πάρα πολύ απλά. Θα εξασφαλίσετε ότι αυτό το νομοθέτημα θα τεθεί σε κίνηση το ταχύτερο δυνατό και θα υποβληθεί από την Κομισιόν. Σας ευχαριστώ. Από τι γνωρίζω εγώ ο ίδιος, υπάρχει μια μελέτη εν εξελίξη για να βρεθεί μια ε, απάντηση στο αν είναι απαραίτητο να υπάρξει μια νομοθεσία για το θέμα αυτό. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι η ευζοία των ζώων είναι ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα και πρέπει να, να τύχει τη σωστή ρύθμιση. Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των επιστημονικών μελετών. Θα τύχει συζήτηση το θέμα αυτό στο Σώμα των Επιτρόπων και το αν θα υπάρξει πρόταση για νέα νομοθεσία, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει από το Σώμα των Επιτρόπων. Η προσωπική μου θέση είναι σαφής. Χρειάζεται να βρεθεί μια λύση, χρειάζεται να επιταχυνθεί η επίλυση αυτών των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Τσούλο, έχετε το λόγο για την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτά που είπατε στην αρχή της παρουσιάσεώς σας. Ε, ξεκινήσατε, λέγατε ότι θέλετε να προστατεύσετε την υγεία των ανθρώπων, θέλετε να προωθήσετε δράσεις για να βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής και την υγεία στη ζωή. Βασιστήκατε στην πρόληψη και την πρόθεση τρόπων ζωής ε, βιώσιμων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω βάσει ενός συγκεκριμένου θέματος ε, των, των κακών τροφίμων, των junk food Αυτά επηρεάζουν και την ευζοία και, οικονομικά επηρεάζουν, διότι μετά απαιτούνται θεραπείες. Καλές οι πρωτοβουλίες για να προωθούν οι υγιεινοί τρόποι ζωής, αλλά κάποιες χώρες ξεπερνούν τα όρια και οθετούν κάποιες δράσεις νομοθετικές για να αποτρέψουν τους ε, πολίτες από το να καταναλώνουν αυτά τα ανθυγινά τρόφιμα. Σας ρωτώ, είσαστε διαθέσιμοι να τοποθετηθείτε τέτοιο το τρόπος και να σας πω ότι υπάρχουν μέτρα και εργαλεία που μπορούν να υιοθετηθούν. Ποια? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η πρόληψη των μη μολυσματικών ασθενειών παίζει ένα σημαντικό ρόλο Μάλλον και η υγεία και η διατροφή παίζουν ε, σημαντικό ρόλο. Η υγιεινή ε, διατροφή και η εκπαίδευση, η παιδεία είναι σημαντική. Θα πρέπει τον υπηαγωγείο να ξεκινά η υγιεινή διατροφή και ο υγιεινό τρόπο ζωή και τη οικογένεια. Διότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίε και συνήθειε και συμπεριφορέ ε, μετά η διαχείριση των κινδύνων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και των σχετικών παραγόντων που δημιουργούν κινδύνους. Η κατάχρηση ενοπνευματοδών, καπνού, η υπερβολική χρήση ζάχαρης. Είναι ζητήματα αυτά. Και τα προγράμματα που βοηθούν τον έλεγχο των ε, παραγόντων κινδύνου είναι κάτι που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να παραπέμπουν σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να προωθήσουν κάποια προγράμματα. Ακόμα και ευρωπαϊκοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων. Μόνο 3% των πόρων αφορούν την πρόληψη και αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα διαθωτικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων πρόληψης. Μπορούμε να τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Χρειαζόμαστε ένα σύμπλεγμα προγραμμάτων που θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, θεσπίσουν ε, κάποια μέτρα, ε, συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη μη μολυσματικών ασθενειών. Ευχαριστώ, συνάδελφος μου είχε το λόγο. Οι πολίτες και οι καταναλωτές στην Ευρώπη συνεχίζουν να αγνοούν εις βάρος της υγείας τους τι τρώνε. Στην Ευρώπη και κυρίως στην Ιταλία εξακολουθούν να μπαίνουν από τρίτες χώρες διάφορα τρόφιμα και παράγωγα μη γενετικών τροπημένων οργανισμών και ζωοτροφές που μολύνουν τα ζώα τα οποία καταλήγουν στο τραπέζι μας. Δεν πιστεύετε ότι η προστασία τη διατροφή των πολιτών πρέπει προβλέπει ένα σύστημα ετικετοθεσία που θα είναι πιο διαφανέ, που θα λαμβάνει υπόψη και στην περίπτωση τυχαίων μολύνσεων και των παραγόγων προϊόντων που προέρχονται από ζωοτροφέ και μη γενετικά τρόφιμα. Μία ετικετοθεσία θα πρέπει. Δεν δείχνει ποιε οι συνέπειε μπορεί να έχουν στην ανθρώπινη υγεία γενετικά τροπημένοι οργανισμοί. Δεν θα πρέπει να αναθεωρηθεί το επίπεδο της μόλυνσης που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 0,1%. Βλέποντας το TTIP, μήπως θα πρέπει να ε, καλυφτούν τα κενά, ούτως ώστε να μην κατακλειστούμε από γενετικά τροπημένους οργανισμούς ανεφ, ε, ελέγχου. Και από ποια επιστημονικά στοιχεία μπορεί να βασιστεί η σιγουριά σας ότι δεν θα υπάρξει αυτή η μόλυνση με γενετικά τροπημένους οργανισμούς. θα συμφωνήσουμε νομίζω όλοι πως ε, το σημαντικότερο εδώ πέρα είναι τα επιστημονικά στοιχεία. Και πρέπει βεβαίως να εμπιστευόμαστε την ανεξαρτησία των ε, στοιχείων αυτών. Αν υπάρχει χρηματοδότηση από τη βιομηχανία τότε μπορεί να υπάρξει κάποια κατάχρηση, όπως παραδείγματος χάρη στην οδηγία του καπνού. Είδαμε δημοσιεύσεις που έλεγαν πως δεν βλάπτει την υγεία, παραδείγματος χάρη. Δεν ήταν επιστημονικά στοιχεία αυτά, ήταν προπαγάνδα σκέτη. Οπότε πρέπει να βασιστούμε σε ανεξάρτητα επιστημονικά στοιχεία, αξιόπιστα, και βεβαίως ε, να... και έχουμε και τον ε, Codex Alimentarius όπου έχουμε κωδικοποιήσει ε, κάποιες απαιτήσει. που βεβαίως βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και πρέπει να εφαρμοστούν. Π.χ. αν έχουμε τρόφιμα χαμηλής ποιότητας πρέπει να δούμε τι συστήματα ελέγχου έχουν τα κράτη-μέλη και τι ε, μπορούν να κάνουν. Αλλά είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα, πρέπει να ληφθούν μέτρα και να δημιουργήσουμε ε, κάποια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, πάντα σε έναν διάλογο με τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τελευταίο γύρο των ερωτήσεων και ξαναγυρνάμε στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ο πρώτος είναι ο συνάδελφος Τανασέσκου που Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Υποψηφία Επίτροπε, κάθε χρόνο 1,3 άτομα κάθε χρόνο πεθαίνουν από φυματίωση. Και ιδίως υπάρχει η μορφή της φυματίωσης που αντέχει <clears throat> στα, στα αντιβιωτικά. Παραμένει η υγειονομική περιθέλψη μέσα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών που δεν έχουν πάντα μπορέσει να αντιμετωπίσουν αυτή τη διαμεθοριακού χαρακτήρα δράση. Είναι απαραίτητε οι κοινέ δράσει Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί αυτή η επιδημία, ιδίω τη στιγμή που το Παγκόσμιο Ταμείο για την Υγεία έχει αποσυρθεί από την Ευρώπη και υπάρχουν ε, πολλοί πιο ακριβά φάρμακα μονάχα για τις νέες μορφές φουμεθίωσης που αντέχει στα αντιβιωτικά και που έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό επιτυχίας. Μόνο ένα στα, στους τρεις θεραπεύεται αποτελεσματικά. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν κύριε Ανδρίου Κάιτης, εσείς ως Επίτροπος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θα αναγνωρίσετε τη φυματίωση ως μια σοβαρή διαμεθοριακή απειλή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάρετε τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει ο έλεγχος αυτής της επιδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Το αν μια ε, ασθένεια είναι επιδημία ή πανδημία, αυτό υπόκειται σε σαφείς κανόνες. Δεν μπορώ εγώ να σας πω τους κανόνες, αυτό είναι θέμα των επιδημολόγων, αλλά πρέπει να μείνουμε πιστοί στους κανόνες αυτούς και να τους σεβαστούμε. Το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες μορφές φυματίωσης που αντέχουν στα αντιβιωτικά, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά από τη μία πλευρά τα εθνικά κράτη μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία των κοινωνικών ομάδων οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες όπως είναι οι τοξικομανείς παραδείγματος χάρη που υπόκειται σε πολύ μεγάλους κινδύνους αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουν τα κράτη-μέλη για τα άτομα τα οποία μπορούν να έχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα υγείας και άτομα τα οποία βρίσκονται σε ε, υποβαθμισμένα κοινωνικά στρώματα. Πρέπει λοιπόν εδώ να υπάρξει καταρχήν μια κοινωνική υποστήριξη, μια βελτίωση της διατροφής των ατόμων αυτών, μια βελτίωση γενικά της υγείας τους. Έχω αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και ως υπουργό στη χώρα μου. Πρέπει όμως να ζητήσουμε και από τα κράτη-μέλη πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το γενικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ένα ιατρικό πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί και από κοινωνική πτυχή και να εξασφαλίσουμε ότι οι πιο ε, <clears throat> εκτεθειμένοι στους κινδύνους αυτούς από μορφές φυματίωσης που αντέχουν στα αντιβιωτικά ότι θα μπορέσουν να τους υποστηρίξουν και να εμποδίσουν την περαιτέρω επέκταση αυτού του προβλήματος. Φυσικά είναι ένα πρόβλημα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το έχει τονίσει ως ένα ιδιαίτερο στοιχείο του προγραμματός τους και εγώ φυσικά θα σας υποστηρίξω απόλυτα στο θέμα αυτό ως Επίτροπος γιατί υπήρξα γιατρός και στο παρελθόν και γνωρίζω ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. Αν θα γίνει πανδημία αυτό είναι κάτι το συζητήσιμο. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γκίζεκ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες ε, προκλήσεις σε ό,τι αφορά τις ε, ε, δαπάνες οι οποίες συνδέονται με το σύστημα αυτό. Μια καλύτερη πληροφόρηση θα μπορούσε να βελτιώσει πολύ περισσότερο την χρήση του συστήματος αυτού από τους ε, ασθενείς. Στον τομέα λοιπόν αυτών της επικοινωνίας και της, της επικοινωνίας και της πληροφόρησης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον ψηφιακό κόσμο. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί λοιπόν και το θέμα της ηλεκτρονικής υγείας εσείς είσαστε έτοιμοι να το κάνετε αυτό και τι θα κάνετε για να εξασφαλίσετε ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παροχής υγειονομικών συμβουλών ε, μπορούν να λειτουργούν με διαλειτουργικό τρόπο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία από τις 10 προτεραιότητες της είναι το ψηφιακό θεματολόγιο. Και εδώ βλέπω και την ηλεκτρονική υγεία ακόμα και την κινητή ηλεκτρονική υγεία. Εδώ έχουμε τεράστιες δυνατότητες συζητήσει με τους επιστήμονες, με, τους, ε, με το βιομηχανικό κλάδο και υπάρχει αυτή η δυνατότητα μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, παραγματικά χάρη, κανείς να στέλνει ένα καρδιογράφημα και να παίρνει τις απαραίτητες, ε, να να απαραίτητε μάλλον τις στο κέντρο αντιμετώπιση ασθενειών ή θεραπείας. Ξέρω ότι υπάρχουν αυτά τα προγράμματα και αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Χάρη στην ε, ε, ελευθερία κυκλοφορίας των ατόμων γίνεται ουσιαστικά ένα επιτακτικό θέμα να μπορεί να λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη. Μπορεί λοιπόν η ψηφιακή Ευρώπη να τεθεί στην υπηρεσία της προστασίας των ασθενών. Υπάρχουν τεράστιες ε, δυνατότητες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πώς επομένως θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη τα σχέδιά τους για την ηλεκτρονική υγεία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ήδη μεταφέρει τη συνταγογράφηση σε ηλεκτρονικό επίπεδο, όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν επίσης και οι δυνατότητες να υπάρχει επικοινωνία σε ηλεκτρονικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν τη δυνατότητα να υπάρχει η διαλειτουργικότητα των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας ώστε να ε, μπορεί να εξασφαλιστεί η καλύτερη αντιμετώπιση των ε, ιατρικών προβλημάτων. Είναι σχεδόν απεριόριστες οι δυνατότητες οι οποίες ανοίγονται με τη χρωσή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για τα θέματα υγείας. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος Κάντενμπαχ έχει το λόγο. Εδώ ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, οι μη μεταδοτικές χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, τα καρδιακά νοσήματα, καρκίνος και ψυχικές διαταραχές είναι ε, νομίζω μαζικότατες, 86% των ε, θανάτων και ένα 80% της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας αντιπροσωπεύουν. Επίσης θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται με τις ανισότητες στην παροχή υγείας. Και βεβαίως εδώ πέρα απαιτείται ε, ισχυρή πολιτική βούληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις νέες πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές η υγεία από ό,τι φαίνεται παίζει έναν δευτερεύοντα ρόλο. Πώς θα συνεισφέρετε εσείς ε, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των χρονίων ασθενειών και να είναι υψηλά στην ε, ατζέντα της ε, Κομισιόν. Πώς θα διασφαλίσετε το ότι οι συστάσεις προς τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα ακολουθηθούν και δεν θα είναι απλά ευχολόγια όπως τα τελευταία χρόνια. Και τέλος, ποιους θεωρείτε εταίρους όσον αφορά τα ζητήματα ενημέρωσης για την υγεία. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως σήμερα χρησιμοποίησα τρεις λέξεις. Πρόληψη, προστασία και προώθηση. Εγώ συχνά όταν ακούω πολιτικούς ε, να μιλάνε θεωρούν πως οι τρεις αυτές λέξεις σημαίνουν το ίδιο. Όχι. Οι τρεις αυτές λέξεις υποκρύπτουν διαφορετικές τεχνικές και μέσα που ε, υλοποιούνται διαφορετικά. Σε γενικές γραμμές εγώ δεν ξέρω ούτε μία κυβέρνηση όπου ο υπουργό Γεωργίας, Δικαιοσύνης, ε, Εκπαίδευσης ή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν έχει σχέση με τα ζητήματα υγείας. Όλοι σκέφτονται πώς μπορούν να μειώσουν τις κοινωνικές διακρίσεις, τις κοινωνικές διαφορές και θέλουν να ελέγχουν τους κινδύνους και να αυξήσουν τους πόρους ε, της υγείας. Οι πόροι της υγείας αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθρωπότητα, πολύ περισσότερο από τις επενδύσεις των τραπεζών. Γι' αυτό ακριβώς όταν ε, κοιτάω και βλέπω αυτές τις 10 δεσμεύσεις είτε αφορούν την ψηφιακή πολιτική, είτε την εργασιακή πολιτική, τις αγορές, σε όλα αυτά υπάρχουν στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία και σας διαβεβαιώ πως εγώ θα προσπαθήσω να πείσω τους συναδέλφους μου να υιοθετήσουν ένα πακέτο μέσων. Είναι πολύ σωστό το ερώτημα που θέτετε. Εάν μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως αυτά τα μέσα και εργαλεία πρέπει να εφαρμοστούν ισότιμα σε όλα τα κράτη-μέλη θα μειώσουμε το κόστος της υγείας γιατί ο κόσμος θα αρρωσταίνει και λιγότερο. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να αντιληφθούμε πως α, πεθαίνει πάρα πολλοί κόσμος πάρα πολύ νωρίς και εγώ θα εργαστώ προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Γκαρντίνη. ένας Γκαρντίνη, και υποψήφια υποψήφια. Επίτροπε, έχω μια ερώτηση. Μπορείτε να δώσετε τον ορισμό σας του ενήμερου και ορίμου καταναλωτή. Όχι με υπόσχεση, ορισμό. Τώρα όσον αφορά τα διατροφικά κριτήρια, τις ενδείξεις διατροφικές και την υγεία, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και θα πρέπει να αποδειχθούν επιστημονικά, θα μπορούν να εμφανίζουν στην ετικέτα μόνο μετά από διοδότηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα επιστημονικά κριτήρια είναι αυστηρότατα κυρίως όσον αφορά την ένδειξη για την υγεία ε, που είναι κάτι που διοργανώνει η Υπηρεσία Τροπίμων, η Ευρωπαϊκή ΕΦΣΑ. Λοιπόν, ε, ζητείτε να κάνει δεξάγει πειράματα τόσο αυστηρά που είναι κάτι αντίστοιχο με αυτά που ζητάμε για τα φάρμακα. Είναι πολύ ακριβό. Πάνω από 500.000 ευρώ κοστίζει κάθε υπόθεση αυτό θα βγάζει εκτός μάχης τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ρωτώ, σκέφτεστε στην αναθεώρηση του κανονισμού το αντιμετωπίσετε αυτό. Διότι διαφορετικά πραγματικά δημιουργούμε την εντύπωση ότι η νομοθεσία για τα τρόφιμα ευρωπαϊκή θα ζημιώσει τους μικρούς παραγωγούς, τις μικρές επιχειρήσεις και πολλούς δικούς μας σημαντικούς εθνικούς ε, παραδοσιακούς ε, παραγωγούς. Ευχαριστώ. Norėčiau pasinaudoti mediko terminą. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω λίγη ιατρική ορολογία για να σας πω ποιος είναι ο ενημερωμένος καταναλωτής. Quantum satis, όπως λέμε στην ιατρική. Έτσι, ωραίο, δεν ακούγεται. Δηλαδή, όση πληροφορία χρειάζεται. βρίσκουμε κάθε φορά την ισορροπία. Ούτε υπερβολική ε, πληροφορία, ούτε ελάχιστη. Αν έχουμε μία ετικέτα με 28 διαφορετικές γλώσσες με ψήρες ε, τα, γράμματα, δεν μπορεί κανείς να το διαβάσει και χρειάζεται μεγεθυντικό φακό έτσι και κάπου χάνεται νομίζω η κοινή λογική. Και δεν μπορούμε μετά να αξιολογήσουμε το προϊόν αντικειμενικά. Οι πληροφορίες δεν αναγκινάνε μόνο τυπωμένες στο χαρτί, υπάρχουν και ηλεκτρονικά μέσα. Ή μπορεί να έχουμε τη διεύθυνση του site πάνω στην ετικέτα. Ε, πολλοί προσπαθούν να μειώσουν, πολλές εταιρείες προσπαθούν να μειώσουν τη χρήση χαρτιού και ακριβώς παραπέμπουν στο site. Και βεβαίω θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να δώσουν την ε, νομική δυνατότητα. Το πρόβλημα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να δούμε τις ε, σύγχρονες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που δίνουν για την ενημέρωση του καταναλωτή για να μην χαθεί ο καταναλωτής. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφε Μπόρζαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Δόκτωρ Αντρικάητης, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε ξανά στην Επιτροπή μας. Ε, αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις σχετικές με την υγεία. Κάποιες από αυτές είναι αυξημένος αριθμός ασθενειών, αυξανόμενος αριθμός των ασθενειών και προβλημάτων όπως είναι η παχυσαρκία που έχει αρνητικές συνέπειες. Ένας από τους βασικούς δείκτες προόδου όσον αφορά την ιατρική με θετικά συνεπακόλουθα είναι η επέκταση του προσδοκίμου ζωής προσθέτουμε περισσότερα ε, χρόνια ζωής. Έχουμε μια δημογραφική αλλαγή. Αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις. Διότι μαζί με τα ιατρικά επιτεύγματα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο πώς χρησιμοποιούμε τα μέσα. Ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτόμαστε και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Ερώτηση. Προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το όλο πρόβλημα της δημογραφικής αλλαγής και της βιωσιμότητας των συστημάτων αγίας, υγείας συγγνώμη, και με ποιο τρόπο. Διότι δεν θα πρέπει να αφήνουμε αυτό το θέμα μόνο σε επίπεδο κάτων μελών. Πιστεύω ότι καλύτερο θα ήταν να το εξετάζουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, εγώ συμφωνώ με απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να αποκομίσουμε μια προσθέμενη αξία. Δεν πρέπει να παραμείνουμε μόνο σε επίπεδο επικουρικότητος. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε βέβαια τις συνθήκες, οι οποίες κάνουν σαφείς διαχωρισμούς αρμοδιοτήτων, γιατί πρέπει να λειτουργήσουμε με βάση πάντα τις συνθήκες, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διαδεσή μας, τη δυνατότητα συντονισμού, μεταλαμβάνευση βελτίστων πρακτικών, και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και τους φραγμούς που υπάρχουν, να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις, σε κοινά κριτήρια για καλύτερη αξιολόγηση των υγειονομικών συστημάτων. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τα κρατημέλη μπορούν να κάνουν και να πάρουν και πρωτοβουλίες με την ενισχυμένη συνεργασία, εφόσον το επιθυμούν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα που δίδεται από τις συνθήκες. Η ενισχυμένη συνεργασία είναι μέσα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε διάφορους τομείς, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν με πιο γρήγορα βήματα προς την επίτευξη υψηλότερου επίπεδου υγειονομικής προστασίας. Γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα μόνο με μια φόρμουλα πρέπει να συνεργαστούμε και ιδίως πρέπει να συνεργαστούμε στα θέματα που έχουν διαμεθοριακό χαρακτήρα. Θυμάμαι τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την, Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Αυτό ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα που δεν πρέπει να την ξεχάσουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για μια ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτό για τις χρόνιες ε, ασθένειες, για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, θα πρέπει μέσα στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να αναζητήσουμε λύσεις για, τις οποίες, για να αντιμετωπίσουμε παραδείγματος τη θεραπεία των ηλικιωμένων στην οικία τους και όχι σε νοσοκομεία και τώρα. Πρόεδρε, η πρόσβαση στην ε, ποιοτική περίθαλψη είναι βασικό δικαίωμα των πολιτών της Ευρωπαϊκής και βασικό ε, στοιχείο των συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής Δεν είναι όμως η πραγματικότητα σήμερα. μείωση ανισοτήτων στον τομέα της υγείας είναι κρισίμου σημασίας για την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής και την υγεία τους θα, θα πρέπει να ληφθούν εστιασμένε δράσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εύκολη, Κυρίω από πρόληψη μέχρι θεραπεία, κυρίω με χρόνιε ασθένειε, με προβλήματα ογκολογικά, σπάνιε ασθένειε, παιδιά, ενήλικε, που είναι σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Θα, θα συμμετάσχουν οι οργανώσεις κοινωνία των πολιτών όπω οργανώσει και σωματεία ασθενών στην προσπάθεια που θα γίνει. Αναφέρατε σαν προτεραιότητα την πρόληψη πρόληψη και σύμφωνα με το κοινωνικό συμφέρον υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα ξεκινήσατε ανεξάρτητη νέα μελέτη για το τι γίνεται με την ακτινοβολία στις συσκευές ε, τηλεπικοινωνίας και μικροκύματα, κυρίως όσον αφορά ασθένειες που σχετίζονται με καρδιαγγειακά και ενδοκρινικά προβλήματα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Αναφερόμενοι στην ανάθεση αυτής της μελέτης σχετικά με την ακτινοβολία, πώς επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία. Εάν η σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου το θέσει το πρόβλημα, εμεί θα πρέπει να αντιδράσουμε. Πρέπει να συμπιστήσω την προσοχή επί της παρούσης καταστάσεως. Χρειάζονται συγκεκριμένα στοιχεία, κάποια συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει να μπούμε και να εξετάσουμε τις λεπτομέρειες όσον αφορά τη θεραπεία ασθενειών, κυρίως σπανίων ασθενειών και ασθενειών παιδικών θα πρέπει να εξετάσουμε την οδηγία για τη δυσυνοριακή περίθαλψη. Έχουμε προβλήματα με τις σπάνιες ασθένειες και καμιά φορά έχουμε φάρμακα που είναι συγκεκριμένα κέντρα και μπορούν τα παιδιά να πάνε για περιθάψη. Έχουμε περιπτώσεις όπου Έχουμε πολύ λίγες ε, περιπτώσεις μια συγκεκριμένη ασθένεια. Είναι πολύ σπάνια. Μπορεί να έχουμε μόλις 12 τέτοιες περιπτώσεις και μπορεί να δούμε αν υπάρχει κάποιο κέντρο που μπορεί να περιθάψει αυτά τα άτομα. Και χρειάζεται και αναλυθεί το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Χρειάζονται κατεπηγόντως λύση αυτά τα θέματα και πρέπει με ενεργό τρόπο να κινηθούμε επιδιώκοντας λύση. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο για τελευταία ερώτηση στη συνάδελφο Μάρετ Μαγκίνες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα κληρονομήσετε πολλούς φακέλους και ένας από αυτούς είναι η αναθεώρηση της ε, νομοθεσίας ιατρικών συσκευών. Και τα ζητήματα ασφάλειας των ασθενών και της καινοτομίας είναι πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο. Πώς βλέπετε την ισορροπία μεταξύ αυτών των ζητημάτων, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας στο μέτωπο αυτό, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος, ειδικά όσον αφορά τις εγκρίσεις ε, των συσκευών αυτών και βεβαίως ε, πόσο σημαντικές είναι οι ιατρικές συσκευές όταν μιλάτε για καλύτερη υγεία για όλους. Για... Τα αν θα μπορούσαμε όλοι σήμερα να φανταστούμε τα εξωτερικά ιατρία, τον οικογενειακό μας γιατρό, χωρίς ιατρικές συσκευές. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει πως οι ιατρικές ε, συσκευές έχουν τεράστια σημασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές όταν μιλάμε για τον εξυγχρονισμό του συστήματος υγείας. Γιατί αν υπάρχει πρόβλημα με τις ιατρικές συσκευές τότε πώς θα στείλει παραδείγματο χάρη ο γιατρός ε, πληροφορίες ε, σε ένα ιατρικό κέντρο όταν βρίσκεται στη Λιθουανία να στείλει τις πληροφορίες σε μια άλλη χώρα. Και αυτό βεβαίως ε, σχετίζεται και με τη βιομηχανία, την καινοτομία, την έξυπνη καινοτομία στον τομέα της υγείας. Γι' αυτό λέω ακριβώς πως ο τομέας της υγείας είναι πολύ ενδιαφέρον. Δημιουργεί πλούτο, ΑΕΠ. Ένα τομέα ε, που μελετάει η Κομισιόν και μετά χρησιμοποιεί τις ε, μελέτες αυτές. Εγώ είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος σε αυτές τις ε, συζητήσεις όταν είχε η Λιθουανία την Προεδρία της Ένωσης και θέλω να ευχαριστήσω τους συγητές ε, της Επιτροπής σας που συνεισέφεραν σημαντικά στην έκθεση Ροτ Μπέρεντ και Πέτρι Λίζε και είδαμε και τις αδυναμίες βεβαίως που υπήρχαν. Βεβαίως έγιναν πολλά τότε στον τομέα αυτών, αλλά θα είναι σημαντικό το ζήτημα αυτό και οπωσδήποτε θα με απασχολήσει. Ευχαριστώ καταρχάς του συναδέλφους για τις ε, ερωτήσεις που έθεσαν και ευχαριστώ τον Επίτροπο για τις απάντησεις που έδωσε. Θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για μια σύντομη ε, παρέμβαση καταληκτική που δεν, θέλουμε, δεν θα θέλαμε να πάνω πέντε λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμο μέλη του Κοινοβουλίου, θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που μου δώσατε να έλθω ενώπιόν σας στο σπίτι των λαών της Ευρώπης. Χαίρομαι που μπορέσαμε να συζητήσουμε θέματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τα θέματα της υγείας και της προστασίας των τροφίμων η Ευρώπη πρέπει να παίξει πρωτοπόρο ρόλο στον κόσμο σε όλους τους τομείς και σε αυτά περιλαμβάνονται και η υγεία, η ασφάλεια των τροφίμων. Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να δείξουμε σε όλο τον κόσμο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα παγκόσμια προβλήματα και τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ως ιστορικός μπορώ να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καλύτερη λύση για να προστατεύσουμε την ανθρωπότητα από τους πολέμους, από το μίσος και άλλες ασθένειες αυτού του είδους. Τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον υγειονομικό τομέα και την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων είναι το καλύτερο παράδειγμα για τον κόσμο μας για να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων. Ως ε, πολιτικός μπορώ να πω ότι όλες οι πολιτικές παρατάξεις είναι ιδιαίτερα ταιριαστές για τις απόψεις τους όταν πρόκειται για τα θέματα της υγείας. Εγώ ως βουλευτής, ως ε, ένα άτομο που έχει σταθεί εκτοπισμένο στο παρελθόν του και έχει επανέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως υποψήφιος επίτροπος, όλα αυτά είναι πολύ συγκινητικά για μένα. Από τότε που ήμουν μικρός από τότε που έτρεχα στην τούντρα της Σιβηρίας ήθελα να φτάσω σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Εντάξει, πιο σοβαρά θέλω να σας πω ότι πάντα ονειρευόμουν ένα διαφορετικό κόσμο, ένα πιο λαμπρό κόσμο όπου θα μπορούσα να βοηθήσω τους ανθρώπους τους συνανθρώπους μου. Αυτό προσπάθησα να κάνω σε όλη μου τη ζωή. Αγαπητοί λοιπόν συνάδελφοι, αν συμφωνήσετε, εγώ θα μπορέσω να αφοσιωθώ ως επίτροπος στους ανθρώπους, στην υγεία τους, στην ευζωμία τους. Ένα πράγμα μπορώ να σας υποσχεθώ, θα εργαστώ σκληρά και θα συνεργαστώ μαζί σας και μαζί όλοι μπορούμε να το επιτύχουμε. Κάτι ακόμα θέλω να τονίσω. Έχουμε εδώ πέρα τη βίβλο μας, τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση το άρθρο 16 στην ένατη παραγραφό του λέει ότι η Προεδρία του Συμβουλίου θα ασκείται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ε, με εναλλαγή σε επίπεδο ισότητας. Δική μου πρόταση ήταν αυτή στη συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης. Όλοι πρέπει να είναι σε επίπεδο ισότητος και όλοι πρέπει εξίσου να αγωνιστούν για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Επίτροπε που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας και που σεβαστήκατε και το χρόνο του πινκ-πονγκ που καμιά φορά είναι πολύ περιορισμένος διότι για κάποια θέματα χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να μπορεί να απαντήσει κανείς. Αυτοί είναι οι κανόνες στους οποίους κινούμεθα και τους κανόνες αυτούς ε, σεβαστήκαμε κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Όπως σημειώσατε κι εσείς, Ανακοινώνω τη συνεδρίαση των συντονιστών θα λάβει χώρα για την αξιολόγηση της ακροάσεως σήμερα ανάμεσα στις 3 και στις 4 το απόγευμα και κάποιοι συντονιστές θα κάνουμε την αξιολόγηση που αφορά την επίδοσή σας σήμερα στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ όλους για μια ακόμη φορά συνεργασία. Ζητώ συγγνώμη που χρησιμοποίησα το σφυράκι σε κάποιες φάσεις ήταν αναγκαίο για να μπορέσουμε να ε, παραμείνουμε εντός των χρονικών ορίων του κανονισμού. Ευχαριστώ και τα ξαναλέμε αργότερα.